Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Κοιτώ το ρολόι μου και η ώρα είναι 9 ε, και 6 λεπτά. Και όχι 8 και 6, κάπου βλέπω γράφει 8 και 6. <laughs> Τι έγινε, νωρί ήρθα. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει η συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Και μου επιτρέπετε ε, να σας ρωτήσω αν θέλετε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Αν υπάρχουν σχόλια μπορεί να εγκριθεί αυτή χωρίς καμία αλλαγή. Δεν βλέπω κανένα να ζητεί το λόγο. Δεν έχω και ανακοινώσεις αυτή τη φορά επιπλέον να σας κάνω. Θα συνεδριάσουν ε, το απόγευμα οι συντονιστές όπου θα έχουμε περισσότερες προφορίες για να σας ανακοινώσουμε αύριο το πρωί. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο τρία της της διάταξης, χρήση της ζώνης συχνοτήτων 470 790 MHz στην Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Το Φεβρουάριο ελήφθη ε, μια απόφαση, σχέδιο απόφασης μάλλον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει αλλαγές στη χρήση των συχνοτήτων, αυτή τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα στα 700 MHz. Ξέρετε ότι ήταν διάσημα το θέμα και πολύ γνωστό. Αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούν ε, ε, τα ραδιοτηλεοπτικά ε, κανάλια, αλλά θα περάσει στην ευρυζωνικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του πακέτου τηλεπικοινωνιών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τόγια και το σχέδιο έκθεσής της θα συζητηθεί στις 27 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρίς έγγραφο. Άρα μόνο βάσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχίζουμε λοιπόν και παρακαλώ την πρώτη αντιπρόεδρό μας, την κυρία Τόγια, να παρουσιάσει τις απόψεις της. Πατρίσια, έχεις το λόγο. Grazie Presidente, lei ha già eh, molto bene inquadrato questo e Πρόεδρε, πολύ καλά τα παρουσιάσατε εισαγωγικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά είναι και πάρα πολύ απλό. Ε, το περιεχόμενο Επίσης ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξη ψηφιακή αγορά, ενιαίας μάλιστα ψηφιακή αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον τελικό στόχο που έχει η Κομισιόν, δηλαδή να δημιουργήσει τις συνθήκες ή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε μια ζώνη όπως εκείνη των 700 που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποιότητος ε, εκπομπής ποιοτικής και έχει και μια μεγάλη σημασία σε κάποιες απομακρυσμένες ζώνες που δεν φτάνουν άλλες συχνότητες. Να την διαθέσουμε λοιπόν για τις υπηρεσίες τις ευρυζωνικές, τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των ε, τηλεπικοινωνιών και των ευρυζωνικών. Είναι σημαντικό και είναι και απλό, γιατί η διάταξη στην ουσία αφορά ή στην προετοιμασία όλων των ενδιάμεσων βημάτων, ώστε από την ημερομηνία που προβλέπει η Κομισιόν το 2020 να έχουμε όλες οι αδειοδοτήσεις της ευρυζωνικής χρήσης για τη ζώνη των 700, το οποίο σημαίνει για κάποιες χώρες κάποιες τροποποίησεις, αλλαγές που μερικές φορές θα είναι και σημαντικής κλίμακας. Η δέσμευση λοιπόν που είναι να χρησιμοποιήσουμε τη ζώνη αυτή των 700 που σημαίνει ότι εκείνες οι υπηρεσίες ε, τηλεπικοινωνιών που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν άλλη ζώνη θα πρέπει να μεταφερθούν. Νομίζω πάντως ότι είναι σημαντικό και γι' αυτό ήθελα να το τονίσω ότι ο τελικός στόχος δηλαδή, της διατάξεως είναι σημαντικός. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή το στόχο αυτό για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που γνωρίζει ότι θα πολλαπλασιαστούν ε, πολλές φορές ε, στα επόμενα δέκα χρόνια η υπηρεσία σε αυτού του χαρακτήρα και της υψηλής τεχνολογίας να δείξει λοιπόν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις υπηρεσίες αυτές. Ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε παγκόσμια. Ώστε να συνοδεύσουμε την ανάπτυξη αυτή γιατί τα ψηφιακά είναι προτεραιότητα για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για όλες τις υπηρεσίες που μας απασχολούν, να αξιοποιήσουμε αυτή την προτεραιότητα. Είναι σημαντικό γιατί διαφορετικά ε, ε, θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις ε, περιπλοκότητες της διατάξεως και όχι στην τελική στόχευση που είναι σημαντική και χρήσιμη. Εάν δηλαδή δεν καταλάβουμε, δεν γίνει κατανοητό γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα δοθεί εντύπωση ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες χωρίς να κάνουμε και κάτι ουσιαστικό. Είναι σημαντικό οικονομικά και είναι και σημαντικό και κοινωνικά, γιατί μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών. Νομίζω ότι είναι το άρθρο 3 μάλιστα που ακριβώς αυτό υπογραμμίζει. Ότι πρέπει να μπορέσουμε να προσφέρουμε ποιοτικέ υπηρεσίες εντός της αγοράς της ψηφιακή. Δεύτερο πράγμα που ήθελα να υπογραμμίσω πέρα από την τελική αυτή στόχευση είναι και το γεγονό και το λέω ε, στους ε, συναδέλφους ότι σήμερα τα πράγματα στα, κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικά για τη χρήση της ζώνης αυτής. Μιλάω για τη χώρα μου που έχει μια ιδιαιτερότητα έντονη έχουμε έντονη χρήση τηλεπικοινωνιών ή στη ζώνη αυτή και επομένως η προσαρμογή στην κοινή αυτή απόφαση θα επιφέρει δυσκολίες, τις οποίες θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί, ούτως πίν. Κάποιες χώρες είναι πιο έτοιμες για την προσαρμογή αυτή, κάποιες λιγότερο. Βεβαίω θα είναι μια κοινή απόφαση, θα πρέπει να ισχύσει για όλου, θα πρέπει να είναι δεσμευτική για όλου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε επομένω και ημερομηνίε ναι τελικές ναι, αυστηρές αλλά που να δίνουν την ε, απαραίτητη ε, μικρή ευελιξία, μικρό περιθώριο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις προσαρμογές που θα χρειαστεί ώστε να μεταφέρουμε από τη μία ζώνη στην άλλη τις υπηρεσίες κτλ. Από το 2017 λοιπόν για τις διασυνοριακές αυτές συμφωνίες που θα αφορά το θέμα για να αποφύγουμε δηλαδή ότι θα υπάρχουν συχνότητες που θα δημιουργούν ε, προβλήματα μεταξύ χωρών και από εκεί πέρα να περάσουμε στην προετοιμασία των αδειοδοτήσεων κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι η ισορροπία μεταξύ της προτάσεως αυτής και της κατάστασης που τελικώς θα έχουμε ως συνομοθέτης για πρόκειται για δεσμευτική απόφαση, συμφωνία, είναι μια κατάσταση win-win. Δηλαδή θα πρέπει να επιτρέψουμε σε όλους τους φορείς των τηλεπικοινωνιών και των ευζωνικών να μπορέσουμε να εξαγάγουν όλες τις ε, ωφέλειες ε, της ανάπτυξης που θα μπορέσουμε επί τη βάση μιας προτάσεως γραπτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. go to the short Και πάμε τώρα στις επόμενες ε, ε, παρουσιάσεις των σχεδόν εισηγητών από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριο Χιόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εισαγωγή της. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα ζητήματα τηλεπικοινωνιών τα οποία εξετάζουμε που δεν αφορούν ουσιαστικά τις τηλεπικοινωνίες. Αλλά το πώς στην πράξη θα καταστήσουμε την Ευρώπη πιο κοινωνική, πώς θα συνδέσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους, πώς θα αξιοποιήσουμε και θα επωφεληθούμε τις Ευρωπαϊκή Ένωσης και πώς θα διασφαλίσουμε ότι η αγορά μας θα είναι κοινωνική και αποτελεσματική ε, και θα εκπληρώνει και ουσιαστικούς στόχους. Όταν ε, γεννήθηκε η πρώτη γενιά τηλεπικοινωνίας, το 3G δηλαδή, ε, η Ευρώπη ετέθευε κεφαλής ήμασταν από τις πρώτες ε, περιοχές που αξιοποιήσαμε στο έπακρο της σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Και είμαστε επικεφαλής και σε πολλές χώρες. Για την τέταρτη γενιά, το 4G, το επόμενο βήμα δηλαδή στην ψηφιοποίηση, εκεί χάσαμε το προβάδισμά μας και είδαμε ότι το προβάδισμα πήρε κυρίως ε, η πλευρά των ΗΠΑ. Και είναι μάλλον ε, παράδοξο πως σήμερα εξετάζουμε πώς θα επηρεάσουμε την επιρροή αυτής της κυριαρχίας. Όμως, Πρόεδρε, εγώ για το 5G, την επόμενη γενιά, την επόμενη εποχή των τηλεπικοινωνιών, θα ήθελα να καταφέρουμε οι συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο το Αμερικανικό να συζητούν πώς θα περιορίσουν το ευρωπαϊκό προβάδισμα. Κανείς δεν θέλει εδώ να πει ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω ως προς την οικονομία. Υπάρχει σοβαρή κρίση στις περισσότερες από τις οικονομίες μας και αυξημένος ανταγωνισμός σε όλες τις οικονομίες μας. Το βορρά μέχρι το νότο, την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Στη σημερινή συζήτηση, μαζί με την εισηγήτρια και τους ε, υπόλοιπους ποιότητες, θα ήθελα να θέσουμε έναν πύχη για να δούμε ακριβώς πώς θα ηγηθούμε της ε, γέννησης της πέμπτης γενιάς. Και ας είμαστε σαφείς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Συμβαίνει ήδη τώρα. Το 4G έχει ήδη εξυγχρονιστεί, περνάει στις επόμενες φάσεις του και τώρα ήδη μπορούμε να δούμε πώς ε, έχουμε φορτηγά χωρίς ε, οδηγούς, χάρη στις νέες τεχνολογίες. Όμως θα υπάρξει και ένα νέο βήμα με την πλήρη εφαρμογή του 5G. Στη ΣΥΠΑ θα ξεκινήσει το 2017. Νότιος Κορέα και αυτη ξεκινούν σιγά σιγά, 2017 και θέλουν το 2020 να υπάρξει πλήρης ε, εφαρμογή. Στην Κίνα το ίδιο, η Ιαπωνία. Στο Ταλίν και στο Κόλμη το έχουμε. Και το, η ζώνη των 700 MHz είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τμήματα της οικονομίας μας θα μπορούν ε, να ε, συνδέονται μεταξύ τους. Ούτως ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία θα τεθεί επικεφαλής ε, και οι επιμέρους κλάδοι της βιομηχανίας και θα κλείσω εδώ, Πρόεδρε. Επομένω, μόνο θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την καθυστέρηση, θα πρέπει να καθυστερήσουμε και σε ό,τι αφορά το ζώνη των 700 MHz. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπασίρ από πλευράς ECR. Ε Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που κάνουμε αυτή την ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την κατανομή φάσματος. Οι Ευρωπαίοι Στρατηγικοί Μεταρρυθμιστέ υποστηρίζουν την ε, ε, στρατηγική για την ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολό τη για να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιούμε στο έπακρον τι τεχνολογικέ εξελίξει για να δώσουμε όθηση στην οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία απασχόληση ε, και τη διατήρηση τη ηγετική θέση τη Ευρώπη στην νέα ψηφιακή επανάσταση. Ω προ το κείμενο, θα ήθελα αρχικά να υπενθυμίσω στου συναδέλφου ότι η κατανομή και διαχείριση του φάσματος αποτελεί βασική προτεραιότητα και αρμοδιότητα των κρατών μελών του ραδιοφάσματος. Ε, και θα πρέπει να τηρηθεί αυτό και το βλέπω ότι συμβαίνει με τα χαρά. Όμως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξει που θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, ω προ το χρονοδιάγραμμα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την καταληκτική ημερομηνία του 2020, η τροποποίηση ε, σε ό,τι αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια προς τις ε, νέες ε, προϋποθέσεις, θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Ήδη έχουν κατανομηθεί 600 εκατομμύρια για αυτό το ζήτημα, όμως θα πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά. Γιατί ορισμένες φορές έχουμε και στήλους έως και 100 μέτρα. Δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει από τη γενέτηρά μου στο Yorkshire. Όμως μπορώ να σας πω ότι πολλά έχουν αναβληθεί εξαιτία των καιρικών συνθήκων. Και υπάρχει περίπτωση και εκεί λοιπόν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν είναι λειτουργούμε μόνοι μας και σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ε, στο κείμενο για να αντικατοπτρίζεται ακριβώς αυτό το ε, θέμα. Στο άρθρο 3 η υποχρέωση των 30 MB ανά ε, δευτερόλεπτο μέχρι το 2020 είναι εξαιρετικά περιοριστικές θεωρώ. Ε, οι διάφορες εφαρμογές και πρότυπα για την κάλυψη του 5G ακόμα εξελίσσονται και έτσι τέτοιες ε, τόσο περιορισμένες διατάξεις μπορούν να αποτρέψουν τους παρόχους να επενδύσουν στο ραδιοφάσμα. Και μάλιστα σε έναν τομέα που έχει τόσο μεγάλες οικονομικές συνέπειες. Περιορίζουμε λοιπόν εδώ του ε, παρόχου να λάβουν υπόψη υποχρεώσει που λαμβάνουν υπόψη γεωγραφικού και άλλου παράγοντε που επηρεάζουν την κάλυψη. Τέλο, δύο λόγια για, το, ε, για τη ζώνη κάτω, κάτω από τα 700 MHz. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι θα χρησιμοποιείται αυτό το φάσμα για τι ε, υπηρεσίε μετάδοση. Όμω, αν έχουμε μόνο το downlink, την καθοδική ζεύξη, αυτό δεν είναι κατάλληλο γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τη σημερινή κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη. Η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση αυτού του ευρωζώνη. Αυτό επιτρέπει και την χρήση white spaces σε κάποια ε, τμήματα του φάσματος ε, που δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν ενδεχομένω να επιτρέψουν τη χρήση εφαρμογών IoT. Αυτό αξιοποιείται από πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αν περιορίσουμε τι υπηρεσίε μόνο στι υπηρεσίε καθοδική έρξης, αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τι δυνατότητε καινοτομία σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κείμενο που λάβαμε από την Ολλανδική Προεδρία, από το Συμβούλιο, ε, το ECR ε, στηρίζει πολλέ από τι τροπολογίε ε, που έχουν ω στόχο να τις κεντάσουν αυτές τι εμφυλάξεις μου. Και προβλέπω σε επικοινωνική συνεργασία με την κυρία Τόγια και του υπόλοιπου κοιόδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους, ε, Ρόντε, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω στα όσα είπε ο συνάδελφος. Νομίζω ότι σχεδόν πέντε χρόνια νωρίτερα είχε συζητηθεί για πρώτη φορά, είχε προταθεί για πρώτη φορά το θέμα αυτό, δεν ήθελε κανείς να μας ακούσει τώρα, τότε. και κατά κάποιον τρόπο είναι κατανοητό γιατί τα UHF χρησιμοποιούνται για τις τηλεοπτικές κυρίως μεταδόσεις και είναι ένα τμήμα του φάσματος εξαιρετικά ελκυστικό. Όμως στο τέλος όλα εξαρτώνται από το περιεχόμενο. Ψυχαγωγία, ενημέρωση, κοινωνικά θέματα, μεταφορές, υγεία, ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό περιεχόμενο εντός της ζώνης και πώς να εξασφαλίσουμε ένα πανευρωπαϊκό πεδίο ανταγωνισμού, να έχουμε διασυνοριακή ε, συμφωνία συντονισμού μέχρι του χρόνου στο τέλος του έτους και να είναι διαθέσιμο για την ε, αποτελεσματική χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό και στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε. Ήδη περιμέναμε, καθυστερήσαμε πέντε χρόνια, ας, ας ε, επιταχύνουμε θα έλεγα. Ευχαριστώ ε, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ραϊμόν από τους Πράσινους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία πράγματα. Πρώτον, εδώ εμείς διαπραγματευόμαστε ε, για ένα πόρο πεπερασμένο που δεν ευρύνεται. Στα ενεργειακά μιλάμε για πεπερασμένους ενεργειακούς πόρους και φυσικούς πόρους, ε, αλλά μπορούμε να ποντάρουμε στις ανανεώσιμες. Εδώ δεν έχουμε ανανεώσιμο φάσμα, ένα είναι το ραδιοφάσμα συγκεκριμένο και περιορισμένο και θα πρέπει να το δεχειριζόμαστε ε, καλά με τεχνολογίες στραμμένες στο μέλλον και να κατανεμηθεί ε, με δίκαιο τρόπο. Δηλαδή να είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν. Έχει δίκιο ο κύριος Ρόντε η κατάσταση πιέζει, επίγει και δεν θα πρέπει να χάσουμε πολλά χρόνια για να καθόμαστε να παρατηρούμε τις εξελίξεις. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, ούτε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Στην παράγραφο 3 γίνεται μια σημαντική αναφορά για συνολική κάλυψη ε, διαδικτύου για όλο τον πληθυσμό. Θα έχουμε πρόβλημα στην πρόσβαση στην αγορά ανάμεσα σε πυκνοκατοικημένε πόλει που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ραδιοσυχνότητε και μπορεί να υπάρξει και μεγάλο κέρδο και στι αεροκατοικημένε περιοχέ που δεν είναι πάρα πολύ ελκυστικό για του παρόχου, γιατί δεν συμφέρει. Εμεί λοιπόν έχουμε την πολιτική ευθύνη να επέμβουμε εκεί και να βρούμε λύσει που να φροντίσουν η αγορά να παρέχει και στις αεροκατοικημένε περιοχέ. Ε, ευρυζωνικότητα. Δεν θα πρέπει η Ήπεθρος να ερημώσει. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο θα αναλάβει η αγορά. Θα πρέπει εμείς να το φροντίσουμε. Ε, γιατί δεν το κάνουν, γιατί δεν τους συμφέρει. Λοιπόν, να μην μπει τώρα αυτή η διαλκυστίδα η πόλη απέναντι στην Ήπεθρο. Αυτό το θεωρώ ως δική μου ε, σημαντική ευθύνη και καθήκον. Οι τεχνολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να εκπέμπει και όχι μόνο να λαμβάνει σήμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με τη δημοκρατία και με την ελεύθερη χρήση και έκφραση στο διαδίκτυο. Χαίρομαι λοιπόν για τις διαπραγματεύσεις, για τις εξελίξεις και τα βλέπω όλα πάρα πολύ θετικά και πολύ επικοδομητικά. much, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα σε όλους τους αδέλφους. Σπανίως έχουμε τη ευκαιρία, μιλάμε εδώ για πολιτισμό στην Επιτροπή μας και επιτρέψτε μου να σας ομολογήσω ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά. Και γιατί αναφέρομαι στον πολιτισμό, γιατί νομίζω θα πρέπει να την έχουμε πάρα πολύ υπόψη μας στην έκθεση αυτή. Το ηλεκτρομαγνητικό ραδιοφάσμα είναι φυσικός πόρος, είναι συλλογικό αγαθό και εμείς έχουμε την ευθύνη να το διαχειριζόμαστε με βάση ε, κριτήρια δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή η ανάπτυξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών να μην θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση των Ευρωπαίων σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Γιατί το λέω, διότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά αλλαγή χρήση του ραδιοφάσματος ε, που σε κάποια σημεία μας φαίνεται πρόωρη αυτή η πρόταση. Δεν αρνούμαστε καθόλου τη σημασία να βοηθήσουμε την καινοτομία στις ψηφιακές υπηρεσίες για την Ευρώπη. Όμως χρειάζεται ένας αφής και ρεαλιστικός οδικός χάρτης που να διαφυλάσει το σημερινό σύστημα παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να διευρυνθεί αυτό το φάσμα πρόσβασης σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικές για τους Ευρωπαίους που δεν έχουν τα χρήματα ή ε, τις τεχνικές δυνατότητες να αλλάξουν ας πούμε δέκτη της τηλεόρασής τους είναι ευρωπαϊκά τα περιεχόμενα, ε, είναι πολλές φορές δημόσιοι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που τα εξασφαλίζουν αυτά και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την προσθέμενη αξία της ίδιας ευρωπαϊκής παραγωγής. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, θα είμαστε στο πλευρό της για να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει ε, την ψηφιακή ανάπτυξη μεν χωρίς να υπονομεύσει τη σημερινή χρήση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών. Είμαστε ναι στραμμένοι προς το μέλλον, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής από την Ιευθυντή, ο κύριος Μορέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Τόια για την πρώτη παρουσίαση αυτή του φακέλου. Θα προσθέσω και εγώ το δικό μου κόκο και το δικό μου σχόλιο στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Οι δικές μας προτεραιότητες εδώ είναι οι εξής. Έχουμε μια θέση υπέρ της επέκτασης ε, στα ευρυζωνικά, αλλά θα πρέπει αυτή η επέκταση να γίνει με μέγιστη διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα ε, και έχοντας υπόψη μας την ανταγωνιστικότητα και τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές που θα χρειαστούν. Ο βασικός στόχος για μας είναι αυτή η, η, ε, η δυνατότητα διασύνδεσης για όλους. Αλλά θα πρέπει να επιτηρήσουμε και να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τη διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε αυτά τα 30 τουλάχιστον μεγαμπίτα ένα δευτερόλεπτο που θεωρεί η Κομισιόν ότι έχει θέσει ο στόχο για το 2020. Εμείς το συμμεριζόμαστε αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικότατα τεχνικά στοιχεία και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η χρήση της ζώνης θα γίνει κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα. Και θα, χρειαστεί να έχουμε ένα, μια συστημική διασύνδεση για όλους τους χρήστες που συνυπάρχουν σε αυτή τη, ζώνη και χρειαζόμαστε ένα σύστημα δημοσίων εκπομπών, δικαιωμάτων, χρειαζόμαστε εξοπλισμό, BMS, χρειαζόμαστε ε, τον προγραμματισμό των ειδικών εκπομπών και εκδηλώσεων. Χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή σε και μια αξιολόγηση αντικτύπου για την εφαρμογή των αποφάσεων και, στην, και την παρακολούθηση που θα εξασφαλίσει ότι οι ωφέλειες της νέας χρήσης της ζώνης θα ξεπεράσουν τις οποιασδήποτε τεχνικές δικαιοσύνες που θα υπάρξουν για τη μετάβαση. Η 30 Ιουνίου του 2022 μας φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξη στόχος για να επιτύχουμε τα 30 MB και θεωρούμε ότι στο άρθρο 5 θα πρέπει να επεκτεθούμε και για τις υποχρεώσεις που, των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 και κλείνω υπογραμμίζοντας ότι για μας είναι τεράστια η σημασία να εξασφαλίσουμε και την έρευνα και η ανάπτυξη που θα χρειαστεί ώστε να επιτύχουμε την αποτελεσματικότητα στην οποία βασίζεται η επιτυχία του όλου της όλης προσπάθειας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Κάπελ από το ομάδα ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα πρόγραμμα ε, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας για να ενισχυθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τρία είναι τα κέντρα βάρους. Πρώτον, το 5G για την κινητή τηλεφωνία, το είπαν ε, οι δύο προλαλήσαντες, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να μην χαθεί και μάλιστα να διατηρήσει την ηγητική της θέση. Δεύτερον, ε, η κεντρική ε, αποθήκευση σε ένα ηλεκτρονικό νέφος iCloud ευρωπαϊκό ε, την ε, ανοιχτή επιστημονική ατζέντα, δηλαδή ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και τώρα υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα και το τρίτο είναι η ασφάλεια ε, στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο. Το όλο εγχείρημα θα κοστίσει 50 δις παρακαλώ από ιδιωτικά και κινητικά κονδύλια. Αλλά σε σχέση με την ψηφιακή εποχή και τεχνολογία και το θέμα που μας απασχολεί δεν έχει να κάνει μόνο η βιομηχανία, ε, είναι η χρήση της ζώνης συχνοτήτων της συγκεκριμένη ε, για την ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη που να καλύπτει όλη την περιφέρεια και την υπεθρο με ευρυζωνική δυνατότητα για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. είναι ιδεώδεις οι συγκεκριμένες συχνότητες, έχουν ευρία κάλυψη και μεγάλη ταχύτητα. Και μάλιστα για τις ε, ασύρματες ε, ε, επικοινωνίες που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από τη τηλεόραση. Η συγκεκριμένη ζώνη 470 με 790 MHz προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί για την ευζωνικότητα, για την τηλεόραση χρησιμοποιείται αυτή τη φορά για την ε, ψηφιακή χερσαία ε, και για τα τηλέφωνα. Υπάρχουν προβλήματα, 13% του πληθυσμού, 65 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από αυτά τα παράσιτα και τις ε, παρεμβολές που γίνονται στις συχνότητες και ιδιαίτερα σε διασυνοριακή εκπομπή και θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχει συντονισμένη διάθεση ε, για ευέλικτη χρήση ε, στη ζώνη κάτω των 700 MHz. Τα λέει όλα αυτά η πρόταση. Το κόστος δεν είναι ευκαταφρόνητο. Ένα ε, 4,2 μέχρι 4,4 δισεκατομμύρια υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μετακυληθεί το κόστος στον τελικό χρήστη που πρέπει να αγοράσει και νέες συσκευές. Ε, θα πρέπει όμως ε, υπάρχει δυνατότητα να είναι ουδέτερες αυτές προς την τεχνολογία. Συν 200 εκατομμύρια, συν κάποια άλλα 890 εκατομμύρια για την ε, προσαρμογή των δικτύων για την ψηφιακή χερσαία τηλεόραση. Τα έσοδα τώρα σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ανέλθουν σε 11 δισεκατομμύρια. Ε, μιλώ πάντα για τη ζώνη των 700. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει και δεσμευτικές ημερομηνίε για την ε, υλοποίηση όλων αυτών, το συντονισμό και το διασυνοριακό μέχρι το τέλος του 2017 και μέχρι τα μέσα του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, προγράμματα τα εθνικά, τα οποία ε, θα τα καταθέσουν μέχρι το χρόνο. Τα δικαιώματα χρήσης θα ε, είναι και μεταβιβάσιμα και εμπορεύσιμα. Και το 2016 ήδη το φθινόπωρο φέτος γίνεται μια παγκόσμια διάσκεψη που θα θέσει τι προδιαγραφέ για το μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για τα σχόλιά σα. Και τώρα προχωρούμε στου υπόλοιπου ομιλητέ. Ο κύριος Μπόνι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ορισμένα σχόλια. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του πακέτου και πλαισίου τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να φύγουμε από την απλή διατήρηση των οδηγιών και να δούμε κάτι διαφορετικό και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό μέσω τη εναρμόνιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απελευθερώσει το Ευρωζώνη σε 700 MHz μέχρι το 2020 σε έναν με έγκαιρο και εναρμονισμένο τρόπο. Δεύτερον, θα πρέπει να δοθεί ε, έμφαση στα κίνητρα για τι ιδιωτικέ επενδύσει. Ε, χρειάζεται απλούστερη νομοθεσία. Πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας ε, και την ποιότητα του διαδικτύου και στο uploading και στο downloading. Ε, είναι πολύ σημαντικός ο ανταγωνισμός, όμως ε, είναι δυσανάλογη η νομοθεσία. Σε κάποιους τομείς πρέπει να δώσουμε κίνητρα για τις επενδύσεις. Ο ανταγωνισμός και οι επενδύσεις δεν λειτουργούν αντιθετικά, αλλά συμβαδίζουν. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι μορφή θα πάρουν. Τέταρτον, χρειαζόμαστε μια πιο εναρμονισμένη πολιτική φάσματο και εναρμονισμένου κανόνε για τον σχεδιασμό κατανομή, ε, χρονοδιάγραμμα κατανομή, ε, προποθέσει αδειοδότηση που θα βοηθήσουν ε, στην αντιμετώπιση του κατακαιρματισμού στην Ευρώπη. Ευελιξία για την χρήση του φάσματο κάτω από τα 700 MHz θα πρέπει να διασφαλιστεί για την εξέλιξη των ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Μετά η αναθεώρηση για το φάσμα των 700 MHz θα πρέπει να γίνει αρκετά νωρί για να προετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή θέση ε, για το WRC23 και έτσι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από το 2025. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Για όλα αυτά θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως είναι η ΜΠΕΡΕΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος με Ευχαριστώ. Ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον του συναδέλφου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο στην αίθουσα που να θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να κάνει τα πάντα ώστε να ηγείται τη τεχνολογία 5G. Ε, Φαίνεται να είναι αυτονόητο. Βέβαια το ζήτημα είναι τον, οι πρακτικές λεπτομέρειες. Πώς θα το κάνουμε. Όπως και οι αντιρρήσεις που θα προκύψουν από κάποια κράτη-μέλη, καθότι αυτή η ζώνη, αυτό το μέρος του φάσματος έχει ήδη δοθεί στα ραδιοτηλεοπτικά. Και βεβαίω δεν θα αναπτύξουμε το σύνολο της οικονομίας μέσω της τηλεόρασης, αλλά θα υπάρξει αντίσταση από κάποια κράτη-μέλη. Γιατί θα υπάρξει κόστος ώστε να, να διανεμηθεί η ζώνη, να έχουμε νέους αποκωδικοποιητές κτλ. Το τηλεοπτικό σήμα εκπέμπεται μέσω διαφόρων συχνοτήτων. Και χρειάζεται μια τεχνολογική λύση ώστε να φτάσει τελικώ στα νοικοκυριά από άλλη ζώνη και αυτό θα χρειαστεί χρήματα. Επομένως, στην προσπάθειά μας να είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης στα 5G το οποίο είναι ένας κοινό στόχος, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις ζώνες για την ανάπτυξη του 5G, αλλά θα πρέπει να βρούμε και μια λογική λύση για τις χώρες εκείνες όπου η ζώνη αυτή μερικώς χρησιμοποιείται ήδη από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Θα πρέπει να βρούμε μια χρηματοδότηση, θα βρούμε τεχνολογικές λύσεις και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Μπλάνκο ε, Λόπεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή αυτή υπογραμμίσαμε την ανάγκη συντονισμού στα θέματα του ραδιοφάσματος και την παρακολούθηση της μετάδοσης δεδομένων για τα κινητά δίκτυα. Εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ώστε να γίνει συντονισμένα η απελευθέρωση της ζώνης των 700 ώστε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα σαφές και να δώσουμε ασφάλεια στους φορείς και στους χρήστες. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία εγείρουν ανησυχίες. Ιδιαίτερα ως προς τον αντίκτυπο που θα έχει στις χώρες εκείνες όπου χρησιμοποιείται έντονα από την χερσαία τηλεόραση η ζώνη αυτή όπως είναι η περίπτωση της Ισπανίας και άλλων χωρών. Χρειάζεται λοιπόν μια αξιολόγηση αντικτύπου από την Κομισιόν που θα έφτανε ω τα 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για, την μετα... για, την... Ε, για τους ε, φορείς που εκπέμπουν τηλεοπτικά και άνω του ενός δις για τους ε, χρήστες, για, για τους πολίτες. Θα χρειαστεί λοιπόν να δούμε να ξαναδούμε μάλλον τον συνολικό αντίκτυπο και το χρονοδιάγραμμα για την συνολική εισαγωγή και μετάβαση της ζώνης αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που συζητούνται εδώ, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου το κυκλοφοριακό στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων αυτή η Επιτροπή ασχολείται με την υψηλή τεχνολογία, με το μέλλον και, τη, και τα ψηφιακά μέσα. Ε, εάν δεν καταλάβουμε εμείς ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, δεν πρόκειται να το καταλαβάλει κανείς. Και υπάρχουν λομπίστες που εκπροσωπούν διάφορα κέντρα που δεν θέλουν να επιταχύνουν και να δουν το μέλλον. Αν αντιλαμβάνομαι τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις εκπομπές και τα λοιπά αλλά το περιεχόμενο, ξέρετε, έχει αλλάξει από τον τρόπο που το κοιτούσαμε στο παρελθόν. Και στη Φιλανδία ο φορέας, ο εθνικός φορέας εκπομπών προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι ηλικιακές κατηγορίες θα έχουν το περιεχόμενο που χρειάζονται. Όχι μόνο ηλικιωμένοι και οι νέοι, όλοι. Και κοιτούν 10 χρόνια μπροστά. Δεν φοβούνται να δώσουν μεγαλύτερο τμήμα κινητή ζώνης Επομένως είναι το περιεχόμενο και ο τρόπος που θα το επιτύχουμε και βεβαίως πρέπει να καλύψουμε και τις τηλεοπτικές ανάγκες αλλά πρέπει να δούμε το τμήμα της ζώνης που εξετάζουμε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Επομένως, θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή εισηγήτρια, η κυρία Τόια έχει ε, υιοθετήσει μια εξαιρετική γραμμή εδώ. Το 5G είναι το μέλλον και ευθυγραμμίζεται και με τα όσα είχαμε συμφωνήσει για την ψηφιακή αγορά. Η εναρμόνιση τώρα για τα 450 είναι σωστή. Είχαμε ήδη συμβαστική πρόταση, πριν από πέντε χρόνια τα είχαμε συζητήσει αυτά δηλαδή. Και όπω λέει και η Κομισιόν, οι χώρε εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση έχουν όρια και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι ε, γειτονικέ περιοχέ. Τώρα οι λεπτομέρειες ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολες. Αυτά, τα όσα έχω ακούσει ήδη από το Συμβούλιο δεν μας αφήνουν να ελπίζουμε ιδιαίτερα. Το Συμβούλιο δεν κοιτάει προς τα εμπρός. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και θα είναι και ο ρόλος της εισηγήτριας για να εξασφαλίσει υποστήριξη. Επίσης το downlink δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τα όσα έχουμε συμφωνήσει διεθνώς. Δεν ξέρω γιατί η Κομισιόν τώρα αυτό λέει. Και τέλος. Η, το Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοτηλεπικοινωνιών θα πρέπει ήδη να προετοιμάσουμε πριν από το 2025 τη θέση της Επιτροπής και της Κομισιόν. Ευχαριστούμε κυρία Κάλλας. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο δεν απαιτείται καμία ευελιξία, είναι οι προθεσμίε. Γιατί η προθεσμία για τον συντονισμό σε ό,τι αφορά την κατανομή του τη ζώνη 700 MHz για την κινητή τηλεφωνία κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά, είπαμε για την ευρωπαϊκή πολιτική για το φάσμα ότι θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κινούνται γρήγορα, αλλά και να τους αποτρέπει να κινούνται αργά. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε τις, ε, την Κίνα και τις ΗΠΑ ε, να τεθούν επικεφαλής, ε, δεν πρέπει να καθυστερούμε. Γι' αυτό και το 2020 ήδη εγώ θεωρώ ότι αποτελεί καθυστέρηση, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχα ορισμένους επισκέπτες από την εκλογική μου περιφέρεια. Είναι εξαιρετική συγκεντρία η Πατρίτσια. Να προσθέσω μόνο τα όσα είπε και η Πέτρα. Όντω, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Βλέπουμε ότι όλα είναι και περισσότερο παρέχονται μέσω ε, κινητών συσκευών. Επομένω, είναι κρίσιμη σημασία όλοι να έχουν αυτή την πρόσβαση και να έχουμε ε, υψηλή ταχύτητα ευρυζωνικά δίκτυα σε όλε τι ε, περιφέρειες για όλου του πολίτε μα, ακόμα και στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ζητεί κανείς άλλος το λόγο. Όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ανδρέας Αγκάης, επικεφαλής μονάδας στην Γενική Διεύθυνση Σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ενθαρρυντικά σχόλια που άκουσα μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ως προς ε, τους ε, στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση. Πρώτον, πράγματι το 2020 είναι σημαντική ημερομηνία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε θέσει αυτή την προθεσμία γιατί εξετάσαμε με μεγάλη προσοχή τα όσα προέκυψαν από την Γενική Διαβούλευση, από τα όσα προέκυψαν από την έκθεση Λαμή ε, και από τα όσα είχαν να πούν όλα τα διαφερόμενα μέρη. Βλέπουμε λοιπόν σημαντικά σχόλια ως προς την ανάπτυξη του 5G, αυτό κατέστησε σαφέ και από τη σημερινή συζήτηση, αλλά και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ηγετική θέση. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν λοιπόν αυτά τα θέματα και να έχουμε κατά νου ότι έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας. Υπάρχει λοιπόν αρκετός χρόνος για να προετοιμαστούμε, για να αλλάξουμε ε, την τεχνολογία και άλλα τέτοια στοιχεία. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα λοιπόν και μπορούν να γίνουν αν αποφασίσουμε γρήγορα και αν αφήσουμε και χρόνο και στον κλάδο να προσαρμοστεί αλλά και στους καταναλωτές χρόνο να προσαρμοστούν σε ό,τι αφορά και την τεχνολογία των εξοπλισμών και το καθεξής. Μετά, για την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και το άρθρο 3 της πρότασης για τις σημαντικές υποχρεώσεις ως προς την κάλυψη. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, θεωρώ. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να αξιοποιήσουμε ε, την ευκαιρία για αυτή τη ζώνη των 700 MHz για να δώσουμε και ένα ισχυρό μήνυμα ως προς τους παρόχους που θα λάβουν ε, αυτό το, ε, αυτή τη ζώνη φάσματος ότι θα καλύψουν και τις περιοχές της υπαίθρου. Θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των προποθέσεων για την αδειοδότηση. Για να υπάρξει εναρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχουμε σαφεί κανόνε ω προ την αδειοδότηση. Να έχουμε λοιπόν συγκεκριμένου στόχου ω προ τα όπως είναι μάλλον τα 30 ΜΜ ένα δευτερόλεπτο. Αλλά όχι μόνο τις περιοχές της Πέθρου, αλλά να καλύπτουμε και το οδικό δίκτυο και το σιδηροδρομικό. Γιατί έχουμε νέες εφαρμογές όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση. Επομένω, πρέπει να τα έχουμε αυτά κατά νου. Γιατί δεν είναι μόνο το να έχει κάποιο ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο όταν οδηγεί ε, στη, στον αυτοκινητόδρομο είναι κρίσιμη σημασία όταν έχουμε την αυτόνομη οδήγηση που εκεί είναι πραγματικά κέριο να υπάρχει σύνδεση με διαδίκτυο. Μετά για, το, για τη ζώνη φάσματο κάτω από τα 700 MHz και τι πρέπει να γίνει με τη μετάβαση. Εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω τη επικαιροποίηση ε, σε νέες τεχνολογίε για να έχουμε αυτή την κατάσταση win-win. Δηλαδή πρόσβαση των κινητών παρόχων στο φάσμα των 700 MHz, αλλά να διατηρήσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά με την ε, διάθεση περαιτέρω φάσματος για τις ε, υπηρεσίες μετάδοσης κάτω από τα 700 MHz. Να συνεχιστούν λοιπόν οι υπηρεσίες που ε, υπάρχουν σήμερα με την επικαιροποίηση σε νέες τεχνολογίες. Εντάξει, αυτό ενέχει κάποιο κόστος, όμως μπορεί να γίνει. για παράδειγμα, θα μπορούμε, μπορεί να αποζημιωθεί το κόστος ε, απόκτησης νέου εξοπλισμού από του καταναλωτέ. Έχουμε τέτοια παραδείγματα όπου η αποζημίωση ε, αυτή για τον νέο εξοπλισμό που παίρνουν οι καταναλωτέ συνάδει με τους ε, κανόνες για τις ε, κρατικές ε, επιχορηγήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτή τη δυνατότητα επικαιροποίηση σε πιο αποτελεσματική χρήση του φάσματος με παράλληλη προσαρμογή της χρήσης σε εθνικό επίπεδο σε ειδικότερες περιστάσεις, γιατί ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την επίγεια ε, μετάδοση περισσότερα από ότι άλλα και εκεί θα μπορούμε να δώσουμε κάποια ευελιξία. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την πρόταση για την ε, εφαρμογή μόνο καθοδικής ζεύξης σε ό,τι αφορά το ασύρματο ευρυζανικό χαμηλών συχνοτήτων. Αυτό συνάδει και με τα όσα ε, αναφέρει η έκθεση Λαμή, η πολιτική ραδιοφάσματος, ή μάλλον η αντίστοιχη επιτροπή για την πολιτική ραδιοφάσματος, Επομένω, ε, μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού περαιτέρω λεπτομέρειες. Θα μείνω εδώ στη διάθεση για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία εισηγήτρια. Καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολύ συνοπτικά θα πω ότι φαίνεται να υπάρχει μια γενική συνένεση, συμφωνία, υπό την έννοια ότι όλοι κατανοούμε τη σημασία της για την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς, για τις ε, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και το υπογραμμίζω εκ νέου για τις πολλές, πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες προς τους πολίτες, για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, μιλήσαμε για μεταφορές, για υγεία, εν πάση τόσο μια γενικότερη χρήση. Επομένως, έχουμε οικονομικές πτυχέ, έχουμε πτυχέ βιομηχανικές, κοινωνικές, τι οποίε αναφέρω τελευταίε, αλλά που είναι υψηλή προτεραιότητας. Όλοι συμμεριζόμαστε λοιπόν το στόχο. Αλλά για να επαναλάβω τις λέξεις του συναδέλφου, υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες στις διάφορες χώρες. Πρέπει να οθήσουμε την Ευρώπη προς την κατεύθυνση και προς το στόχο που θέλουμε με αποφασιστικότητα και θα πρέπει να δώσουμε και τα μέσα στη διάθεση των χωρών και τον χρόνο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ε, τεχνικές δυσκολίες. Έτσι υποχρεωτικά κάποιες χώρε είναι πιο έτοιμες από άλλες, κάποιες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, κάποιες θα καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Για κάποιες χώρε αυτή η ζώνη είναι ήδη υπερχρησιμοποιημένη, δεν έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, χρειάζονται λίγο περισσότερο χώρο. Και επομένως οι διαδικασίες όχι μόνο μεταφοράς χρήσης, αλλά και προσαρμογής ε, και σύζευξης με άλλες ζώνες που θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιες υπηρεσίες ή κάποιες εκπομπές κτλ. Υπάρχει και η δημοκρατικότητα αν θέλετε του περιεχόμενου και της εκπομπής, η χρυσή ισορροπία θα πρέπει να βρεθεί, η διαφάνεια που ανέφερε κάποιος συνάδελφος είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να αξιοποιούμε την ε, χρήση των ζωνών μέσω διαγωνισμών με διαφάνεια, ισότιμα, δίκαια. Και η διατάξη του άρθρου 3 που το, το είχα αναφέρει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι το επανέλαβαν, δηλαδή το θέμα της ποιότητος, της ταχύτητος και της ε, ε, δυνατότητας εκπομπής και διείσδυσης σε όλο το έδαφος είναι ε, πολύ σημαντικό. Θα, αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους πάντοτε. Η διάχυση είναι ε, αυτό που ανταποκρίνεται και στη σημασία του, αυτού που αποκαλούμε κοινωνική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε κάπως διαφοροποιημένες ευαισθησίες, κάποιοι άλλοι βλέπουν περισσότερο τα πολιτιστικά θέματα, κάποιοι άλλοι περισσότερο τα τεχνολογικά. Εν πάση περιπτώσει έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας για να βρούμε μια σωστή ισορροπημένη λύση. Να πω κάτι προς την Κομισιόν, πολλοί το υπογράμμισαν. Ο τεχνικός, τεχνολογικός αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός. Αν χρειαζόμαστε πιο περίπλοκες προσαρμογές που θα έχουν αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις είτε στις ραδιοτηλεπικοινωνίες είτε σε κάποιον άλλο τομέα αυτό έχει σχέση με τον εξοπλισμό του και με τη δουλειά που κάνουν. Όταν όμω μιλούμε για τεχνική, τεχνολογική προσαρμογή που θα πρέπει να επιβαρύνει του πολίτε, είναι διαφορετικό θέμα. Γιατί λέμε ότι όλοι θα πρέπει να αλλάξουν συσκευέ, θα πρέπει να αλλάξουν εξοπλισμό κτλ. Και ε, το αναφέρω σχετικά με το σχόλιο που ακούσαμε για τα κινητά μέσα. Μερικοί λένε πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Μερικοί λένε όχι, χρειαζόμαστε νέε πλατφόρμε, ε, νέου ε, αποκωδικοποιητέ τέλο πάντων. Επομένως, εγώ θα ήθελα να ακούσω μια ουδέτερη αντικειμενική φωνή, αν θέλετε, της Επιτροπής, χωρίς υπεραπλωστεύσεις, και καλό την Κομισιόν. Παρακαλώ πείστε μας τι σημαίνει κόστος. Κόστος για τους χρήστες και κόστος για τις επιχειρήσεις. Με διαφοροποιημένη προσέγγιση. Είμαι σίγουρη ότι μαζί με τους κοιόδες και όλου τους συναδέλφους που θα θέλουν να συνεισφέρουν θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου για την ομιλία αυτή. Λοιπόν, έχουμε τώρα τα εξή. Έχουμε ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα. 27 Ιουνίου είναι για την κατάθεση του σχεδίου γνωμοδότησης. Σε δύο μήνες από τώρα προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 30 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι τροπολογίες θα συζητηθούν στην Επιτροπή μας την 5η Σεπτεμβρίου και θα ψηφιστούν στις 13 Οκτωβρίου, πάντα εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Τον Οκτώβριο δηλαδή είναι η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι η κυρία Τόγια. Και όλους τους σκιώδες και τους λοιπούς συναδέλφους της Επιτροπής μας που έλαβαν το λόγο. Λοιπόν, Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είναι ακριβώς 10 η ώρα. Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Είναι ένα σχέδιο κανονισμού που εντάσσεται στο λεγόμενο πακέτο για την ενεργειακή ασφάλεια που ενέκρινε 16 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δέσμη αυτή προβλέπει μια σειρά μέτρων για να ενισχύσει την αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διατραχές και διακοπές παροχής φυσικού αερίου. Στόχος και δύο κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα προετοιμαστούν καταλήλως έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ε, τις ε, επιπτώσεις της έλλειψης φυσικού αερίου όταν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες περιστάσεις, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ή ε, διακοπές στην παροχή. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, που είναι κάποιος Μπούζεκ. Μου δίνω λοιπόν πέντε λεπτά. You Όπως δίνω σε όλους τους εισηγητές και θα προσπαθήσω να τα χωρέσω αυτά που έχω να πω σε πέντε λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πώς φανταζόμαστε την ασφάλεια, την ενεργειακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έχει αλλάξει πολύ τι τελευταίε δεκαετίες μπορούμε να πούμε χάρη στην κρίση που γνωρίσαμε το 2006 και το 2009. Ξέρουμε όλοι ποια είναι τα αποτελέσματα και των δύο κρίσεων. Και αλλάξαμε την προσέγγιση μας από εθνική σε περιφερειακή και συνέχεια σε ευρωπαϊκή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε αυτή την εξέλιξη, γιατί είναι μονόδρομος. Ε, δεν μπορούμε παρά να το υποστηρίξουμε αυτό. Ο τελευταίος κανονισμός για την ασφάλεια παροχής φυσικού αερίου κατατέθηκε το 2010 και συζητήθηκε πάρα πολύ εντατικά εδώ στην Επιτροπή μας. Θυμάστε, ήταν ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας, Αλέχο, από την Ισπανία. Η οδηγία που προϋπήρχε έγινε τώρα δεσμευτική νομοθεσία και είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα αυτή και ευρωπαϊκή και ενωσιακή. Είναι πολύ σημαντικό. Βίπτει ε, στο άρθρο 194 της Συνδίκης Λισαβόνας που ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Το τονίζω αυτό. Και δεύτερον, ε, συνθέτει ένα ενεργειακό μείγμα. Το κάθε κράτος τα Αυτό παραμένει λοιπόν εθνική αρμοδιότητα, αλλά ευρωπαϊκή επίσης υπάρχει. Ο κανονισμός βελτίωσε πάρα πολύ την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να έρθουν ακόμα εμπόδια και φραγμοί μεταξύ κρατών μελών, να μειωθεί το κόστος. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη διαφάνεια κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια καλή ε, ε, πρόταση και απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Τώρα, πώς βλέπω τώρα ε, τι έχει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να ενισχύσουμε την νομοθεσία του 2010 και τα εργαλεία που έχουμε για να αντιμετωπίζουμε κρίσεις να τα χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σημαίνει αυτό λοιπόν πρόληψη κρίσεων και ε, να προβλέψουμε από πού προέρχονται οι κρίσεις. Για μένα η πρόληψη των κρίσεων είναι πολύ σημαντική για να ε, μην έχουμε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία και θέλω να φέρω τα εξή. Πρώτον, περιφερειακές λύσεις που να βασίζονται σε ουσιαστικά και αποτελεσματικά εθνικά μέτρα φυσικά. Δεύτερον, αλληλεγγύη. Αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας, αλλά ε, κανόνας της εσχάτης διαφυγής, της διαφυγής. Διότι κάθε κράτος θα πρέπει να κάνει πρώτα αυτά που του αναλογούν. Να μπορεί να αντέχει στην κρίση, να διαφοροποιεί τις πηγές, ε, τους προμηθευτές και ε, τους δρόμους, τις οδούς. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι είναι κανόνας η αλληλεγγύη, αλλά όταν κάθε κράτος έχει κάνει τα δικά του πρώτα. Τρίτον, θέλουμε διαφανείς κανόνες ελεύθερης αγοράς στο εμπόριο, το ενεργειακό. Τέταρτον, ε, να δούμε τους γειτονέ μας τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων που είναι μέλη της ε, Ενεργειακής Ένωσης και έχουν δεσμευτεί να τα υλοποιήσουν και να υιοθετήσουν όλα αυτά τα μέτρα. Και το πέμπτο που θέλω να τονίσω είναι συντονισμένες αγορές φυσικού αερίου, να κάνουμε συλλογική αγορά δηλαδή, ε, προμήθεια. Και υπάρχουν και πολύ σημαντικές λεπτομερείς ερωτήσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια ερώτηση ο τρόπο με την οποία τη διατυπώνει. Πιο σημαντική είναι αυτή από την απάντηση. Λοιπόν, ερωτήσει. Χρειάζονται κάποιοι ορισμοί. Παράδειγμα, μέχρι πού θα προχωρήσει η εναρμόνιση των ορισμών του προστατευμένου ε, πελάτη, συμπεριλαμβανομένου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερη ερώτηση, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε μια περιφερειακή ε, υιοθέτηση της αλληλεγγύης. Τρίτον, ε, υποδομές και πρότυπα σε επίπεδο κρατών ή σε επίπεδο ολοκλήρων περιφερειών. Τέταρτον, πρότυπα και προδιαγραφές για τις προμήθειες η δίκαιη μεταχείριση όλων των προμηθευτών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε και να μας προβληματίσουν. Πέντε, ε, εκτίμηση κινδύνου. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι αυτό γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό και πώς ευθυγραμμίζονται και προσαρμόζονται τα εθνικά και τα περιφερειακά σχέδια. Ε, ε, σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ποιος τα καταρτίζει, ποιος τα αναθεωρεί και σε ποιο επίπεδο. Αυτά όλα θα πρέπει να ορίζονται σαφέστατα και με ακρίβεια. Έκτακτε Έκτακτες καταστάσεις, πώς αντιδρούμε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τελευταίο πώς θα εξασφαλίζουμε αρκετή για ε, επαρκή διαφάνεια σε συμβόλαια και συμφωνίες ε, προστατεύοντας ε, τον ανταγωνισμό βεβαίως και την ελεύθερη αγορά και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και κανόνες που ισχύουν. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πολύ εντατική συζήτηση και στο τέλος της συζήτησης έχω το προνόμιο να κλείσω. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο εισηγητής. Πρώτος κοιόδης, πρώτη μάλλον, η κυρία Γκρίφιν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα αυτή που εργάζομαι ακριβώ στην αναθεώρηση της ε, ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο από πλευρά σοσιαλιστών και δημοκρατών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεργάζομαι με έναν τόσο εξαιρετικό εισηγητή όσο ο κύριος Μπουζέκ. Εξετάζοντα τέτοιο ζήτημα όπω είναι η ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη ένα σημαντικό δείκτη σε ό,τι αφορά το συντελεστή εξάρτηση ε, σε εισαγωγές ε, φυσικού αερίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ο συντελεστής ήταν 65% το 2013. Το 95% ήταν 43% και 42% πιο νωρίς. Αυτό σημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτάρκης. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε συγκεκριμένες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να ξεπεράσουμε αυτή την εξάρτηση. Είναι σημαντικό, ιδίω γιατί πρόκειται για μια πολιτική και για στρατηγική πρόκληση που θα επηρεάσει και το μέλλον της Ένωσή μα. Μία πρώτη απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση τη ασφάλεια εφοδιασμού στο φυσικό αέριο και τον σχετικό κανονισμό. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση ε, του υφιστάμενου σχεδιασμού που είναι ανεπαρκής γιατί οι εθνικές πολιτικές δεν λαμβάνουν υπόψη ε, την κατάσταση ως προς την ασφάλεια φοδιασμού σε γειτονικέ χώρες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ανάπτυξη ενός, ε, μιας πιο ολοκληρωμένης περιφερειακής προσέγγισης, ενίσχυση της ε, διάταξης αλληλεγγύης για την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων, όπως ανέφερε και ο Τζέρσι, και εφαρμογή επιπρόσθετων ε, μέτρων διαφάνειας για συγκεκριμένες συμβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια φοδιασμού σε φυσικό αέριο. Εγώ στηρίζω το πνεύμα και των τριών πυλώνων αυτών και εγώ είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς περισσότερη συνεργασία και θα είμαστε πιο δυνατοί στο βαθμό ε, που θα συνεργαζόμαστε και σε επίπεδο κρατών μελών. Προσβλέπω σε ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή και του υπόλοιπου χειώδει για αυτέ τι τρει προτάσει. Όμω, από την άλλη, απογοητεύουμε που η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει καμία πρόταση για την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, που σε τελική ανάλυση είναι το κύριο στοιχείο σε ό,τι αφορά και τους ε, φτωχούς ενεργειακά πολίτες. Το πρώτο αφορά λοιπόν την ενεργειακή πρόκληση και την επένδυση στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα, στην ε, θέρμανση και ψήξη. Νομίζω η στρατηγική για το φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει ε, να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης σε κοινό και στρατηγικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη και την ε, απεξάρτηση από ε, τον άνθρακα. Επίσης, θεωρώ ότι ε, ο διπλασιασμός της ικανότητας του Nord Stream αντιβαίνει στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το, και στις προτεραιότητες ως προς την ενεργειακή ασφάλεια. Η ενέργεια, συνάδελφοι, δεν είναι εμπόρευμα, είναι βασικό κοινωνικό δικαίωμα με ισχυρή πολιτική διάσταση και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και από τις επιχειρήσεις, γιατί και αυτές έχουν ευθύνη για την ασφάλεια φοδιασμού στην Ευρώπη και για όλους ε, τους πολίτες μας ε, στο σύνολό τους. Ε, πραγματικά προβλέπω συνεργασία μαζί σας κύριε Βούσεκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσέσεκ είναι επόμενος ασχιώδης συζητητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αν εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί Όμω, νομίζω ότι βασικό στόχο θα πρέπει να είναι η ενίσχυση τη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ τα ενεργειακά ζητήματα. Κάποια ζητήματα σίγουρα χρήζουν ε, μεγαλύτερης επεξεργασίας, όπως ε, οι ορισμοί και τα κριτήρια που θα μας ε, επιτρέψουν να, να δοθούν μεγαλύτερες εξουσίες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την αξιολόγηση κάποιων συμβάσεων. Προτείνονται ορισμένα κριτήρια, όπως αυτό το 40% που εδώ είναι μάλλον ακαθόδη ζητήματα, όμως θα έχουμε κατά την δυνατότητα να επανεξετάσουμε αυτά τα κριτήρια. Έχουμε την ιδέα της περιφερειοποίησης και της ρήτρας αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος ήδη ανέφερε την ε, αρχή της αλληλεγγύης στην παρουσίασή του, όμως αυτό σημαίνει βέβαια ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, προτείνει συγκεκριμένε διατυπώσεις για να λάβουν υπόψη να ληφθούν υπόψη αυτές ε, οι πτυχές. Αυτό ακούσαμε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ε, και των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ε, την ασφάλεια φοδιασμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί και στην δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια και όλα αυτά θα πρέπει να διευθυνθούν με τον κατάλληλο τρόπο για να διασφαλίσουμε ακριβώς αυτήν την ελληνική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσέσακ. Εξ ονόματος του ECR πήρατε το λόγο. Ο κύριος Τελίτσκα έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Και από πλευρά φιλελευθέρων θα θέλαμε να πούμε ότι η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει βεβαίως να θεωρηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής και να την εξετάσουμε με αμερόληπτο ε, και αντικειμενικό τρόπο για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Ε, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Γκρίφιν περίπου, ότι εξετάσουμε ένα προσχέδιο που ένα από τα κύρια στοιχεία του είναι η αλληλεγγύη. Επίσης έχει ως στόχο μία αποτελεσματική προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε έναν ε, σημαντικό διαχωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως προς το Nord Stream 2. Δεν θέλω τώρα ε, να επεκταθώ παρετέρω, όμως θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε αυτό, ότι η αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το δεδομένο. Επομένως, για να υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη, ε, δεν πρέπει να κινηθούμε παρορμητικά. Θα πρέπει ε, να το εξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή, να βρούμε δικλείδε ασφαλεία και αυτό είναι το πρώτο μου σημείο. Δεν είμαι βέβαιο ότι υπάρχουν τέτοιε δικλείδε ασφαλείας στο κείμενο. Ούτω ώστε κάθε φορά ε, που θα υπάρχει ένα τέτοιο εθνικό συμφέρον και κατακαιρματισμός να μπορούμε να αποτρέψουμε την κατάσταση. Δεύτερον, κάτι άλλο που δεν υπάρχει στο προσχέδιο. Ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Εντάξει, όλοι κατανοούμε περί τίνος πρόκειται. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Όμως, κύριο ζήτημα εδώ, σε αυτό το κείμενο, είναι η ενεργειακή απόδοση και δεν αναφέρεται. Τρίτον, θα είναι ένα αμφιλεγόμενο κείμενο. Με δυσκολία θα περάσει και από το Συμβούλιο. Ήδη ξέρουμε ότι κάποια κρατημέλη αντιτίθενται. Ορισμένα μάλιστα τέτοια κρατημέλη έχουν ιδιαίτερη σημασία ως προς τις περιφέρειες Επομένως, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, για παράδειγμα στην περιφερειακή συνεργασία, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό το κείμενο αποτελεί ένα καλό εργαλείο για να ξεφύγουμε από το διέξοδο. Και τώρα κάτι άλλο. Εγώ είμαι υπέρμαχο της περιφερειακή προσέγγισης, όμως εδώ δεν έχουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση, γιατί μπορεί να υπάρξει και κρίση που θα είναι πολύ πιο σημαντική και οι περιφέρειες να μην μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και ενώ, ας πούμε, στο άρθρο 6 προβλέπεται τι γίνεται σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι περιφερειακοί οργανισμοί, παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γι' αυτό σίγουρα θα πρέπει να λεφθεί υπόψη. Τέλος, δεν έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι έχουμε πραγματικά ένα πλαίσιο εδώ. Είναι ένα σύνολο επιμέρους διατάξεων και μέτρων, όμως δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο, ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω εδώ, αλλά κάποια στιγμή στη συνέχεια σίγουρα θα το κάνω. Και τελευταία παρατήρηση, συνάδελφοι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε αποζημιώσεις. Εάν εφαρμοστεί, ας πούμε, η αρχή της αλληλεγγύης, με σχετικές διατάξεις, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μιλούμε και για ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις, συμπράξεις δημοσίου, ιδιωτικού τομέα. Και, και εδώ πέρα δεν υπάρχει λεπτομερής αναφορά σε εργαλεία αποζημιώσεων για τυχόν ε, επιπλοκές και τυχόν οικονομικές συνέπειες που θα επομιστεί ο ιδιωτικός ε, τομέας. Θα μείνω εδώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με πολλές από τις αρχές που αναφέρατε στην αρχή και θα συνεργαστούμε περαιτέρω στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τούρμας έχει τώρα το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα είμαστε μια πολύ καλή ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την καθοδήγηση του Πρόεδρου. Στην Ενεργειακή Ένωση έχουμε δύο στοιχεία. Αλληλεγγύη και περιφερειακή προσέγγιση. και πρέπει ε, μάλιστα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρόιελ όπου το 2010 στη δική του γνωμοδότηση το συζήτησε το θέμα τοποθέτησε στο κέντρο του ζητήματος την περιφερειακή διάσταση δηλαδή. Η πρόταση Κομισιόν είναι καλή. Και συγχαίρω την Κομισιόν ιδιαίτερα για το παράρτημα 1 που είχε το πολιτικό θάρρος να το κάνει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που αντιτίθενται στο παράρτημα 1. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα. Η Γερμανία δεν ικανοποιείται που είναι σε ομάδα με την Πολωνία και την Τσεχία. Αλλά ζητώ συγγνώμη. Τα <clears throat> χερσαία αυτά σύνορα έχουν σχέση με τον εφοδιασμό, με την αποθήκευση, με τη διαχείριση της ροής του φυσικού αερίου. Πώ θα επιλύσουμε τα προβλήματα αν δεν υποχρεώσουμε τι κυβερνήσει να συνεργαστούν. Η Γαλλία δεν θέλει να είναι στην ομάδα με την Ισπανία. Αλλά και πάλι ζητώ συγγνώμη, αν θέλουμε το δυναμικό να μπορούμε να το διαχειριστούμε και τη ροή να την επιλύσουμε, να είναι ομαλή δηλαδή, και πάλι πρέπει να υποχρεώσουμε τη Γαλλία και την Ισπανία να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεργαστούν. Ελπίζω λοιπόν ότι εμεί, ω Κοινοβούλιο και εμεί ω Επιτροπή στο παράρτημα 1 θα συμφωνήσουμε γιατί είναι μια σωστή προσέγγιση. Πού μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Η προστασία των καταναλωτών και νομίζω ότι ο κύριος Μπούζεκ έχει δίκιο. Ο ορισμός αυτός εκεί δεν είναι αρκετά σαφής. Θα μπορούσαμε ίσως να επιτύχουμε κάτι σαφέστερο εκεί. Η κυρία Γκρίφιν ε, έχει δίκιο και ο κύριος Τίλιτσκα σχετικά με την ε, αποτελεσματικότητα που λείπει ως διάσταση θα ήταν λάθος να μην ενσωματώσουμε στην ασφάλεια εφοδιασμού τα μέτρα αποτελεσματικότητας που μπορούν να ληφθούν για να επικαιροποιήσουμε τον εξοπλισμό και την κατανάλωση των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Επίσης θα μπορούσαμε να βασιστούμε στη βιομάζα διότι το μέλλον του φυσικού αερίου θα είναι να πάμε απευθείας στους αγωγούς και να το χρησιμοποιήσουμε ως πράσινο φυσικό αέριο εντός οικών. Όπως και για τους ε, γεωργούς που δυσκολεύονται με την τιμή του γάλακτος και του κρέατος, πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια της βιομάζας ή στην έννοια του φυσικού αερίου. Και κοιτώντας σε ανατολικές χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, έχουμε πολύ σημαντική γεωργική διάσταση που θα πρέπει να ενσωματωθεί και θα κλείσω. Α, και κύριε Τηλίσκα, έχετε δίκιο. Ίσως να πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί σε κάποιες λεπτομέρειες και πιο συγκεκριμένοι. Και πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα, κάποιες πτυχές ε, αντιστάθμισης. Πρέπει να το διαφημίσουμε αυτό. Θα κλείσω λοιπόν με δύο παρατηρήσεις, ερωτήσεις μία προς την Ολλανδική Προεδρία. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπο της Ολλανδικής Προεδρίας εδώ. Έχουμε. Είναι περίεργο όμως. Γιατί ξέρω τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Ε, υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ των χωρών. Τέλος πάντων. Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ενωμένο Βασίλειο και Ολλανδία για παράδειγμα έχουν μια συμμαχία Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αν θέλετε, μου επιτρέπετε να κλείσω. Αυτό που σημαίνει Συμβουλίο είναι ότι η Ολλανδική Προεδρία έχει προσφέρει την απόσυρση του παρατήματο 1 στη συμμαχία αυτή. Ο κύριο Μπενίτο Ζιλουάγκα από την ΚΟΕ. Και νομίζω ότι εδώ η τελική ευθύνη θα είναι υπό την Σλοβακική Προεδρία ο κύριο Μπενίτο Ζουλουάγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους. Είδαμε την πρόταση κανονισμού και από τη δική μας σκοπιά χρησιμοποιεί τα ίδια φαύλα επιχειρήματα με την ολόκληρη ενεργειακή στρατηγική. Μιλούμε για ασφάλεια στην προμήθεια και για κυριαρχία ενεργειακή. Αυτό τι σημαίνει. Αυτά είναι φρούδες ελπίδες. Τι γίνεται με την εσωτερική κυριαρχία και με την εσωτερική παραγωγή, θα καταλήξουμε στην υδρορογμάτωση. Πάντα θα έχουμε εξάρτηση, μεγαλύτερη ή μικρότερη ασφάλεια, εφοδιασμό, αλλά τελικά εξάρτηση θα παραμείνει παρουσιάζεται στην κοινωνία πιο καθαρό κάψιμο το φυσικό αέριο από τον άνθρακα ή το πετρέλαιο και είναι γεγονός ότι εκπέμπεται λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από την καύση του. Αλλά από τις διαφυγές μεθανίου ε, έχουμε δει ότι ε, υπάρχει πρόβλημα και το μεθάνιο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 86 φορές μεγαλύτερη από το διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν σε δύο θέματα. Πρώτον, τη γεωστρατηγική της ενεργειακής ασφάλειας. Καμιά φορά αυτό μας οδηγεί να κάνουμε συμμαχίες με... Ε, αυταρχικά καθεστώτα και ηγέτες που χρησιμοποιούν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουν τη δική τους ε, θέση και είμαστε με δεμένα τα χέρια μετά όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Η ενεργειακή λοιπόν ασφάλεια έχει και αυτό το στοιχείο της παγκόσμιας ευθύνης και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Και ένα δεύτερο και τελειώνω. Η πρόταση αφήνει στα χέρια της αγοράς ε, το θέμα της κάλυψης ε, καταστάσεων όταν έχουμε έλλειψη ή προβλήματα και ανασφάλεια. Δεν πρόκειται η αγορά να βρει την καλύτερη λύση ούτε την πιο αλληλέγγυα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά θα ψάξει να βρει τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Άρα δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να αφήσουμε στα χέρια ολιγοπολίων και ε, πολυεθνικών που ήδη ελέγχουν την κατάσταση την επίλυση εκτάκτων καταστάσεων και επιγουσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ενεργειακά. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Ευχαριστώ. Η κυρία Κάπελ από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον πρόεδρο δηλαδή. Ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά ε, που λέτε για το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περιφερειακή λύση, για την αλληλεγγύη, για τη ρύθμιση των αγορών με διαφάνεια, τη συμπερίληψη των γειτονικών χωρών και τη συντονισμένη αγορά, προμήθεια δηλαδή ε, φυσικού αερίου. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η πρόταση κανονισμού προβλέπει μεγαλύτερο συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο και καθορισμό συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, περιφερειακή λοιπόν ε, ε, προσέγγιση χρειάζεται και για τη ροή συντονισμός και ασφάλεια εφοδιασμού έχω συγκεκριμένες προτάσεις και εγώ στο σημείο 1 για τον ορισμό των περιφερειών για την αρχή της αλληλεγγύης και να μπορέσει να εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι σαφείς οι περιφέρειες και ισορροπημένες. Εγώ ξέρετε καταγόμαι από την Αυστρία και τώρα έχει μπει σε μια περιφέρεια στο σχέδιο κανονισμού που αποκόπτεται από τις δύο σημαντικότερες χώρες που εισάγουμε που είναι η Γερμανία και η Σλοβακία. Οπότε έχει νόημα τώρα και είναι απαραίτητο στον καθορισμό των ε, περιφερειών να επικρατεί ευελιξία και να υπάρχει ισχυρός διμερής συντονισμός. Να λαμβάνεται υπόψη. Αυτό φαίνεται από το παράδειγμα της Αυστρίας. Μπορεί μια χώρα να συμμετέχει σε δύο περιφέρειες, το έχει και δίπορτο ή δεν ξέρω κάπως να οριστούν καλύτερα οι περιφέρειες. Το ίδιο ισχύει και για τις προδιαγραφές των υποδομών. Τα είπατε και εσείς κύριε Γησίγητα, ε, Ο σημερινός καθορισμός των ε, περιφερειών ε, ε, οδηγεί σε προβλήματα γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και δεν συμπίπτουν οι προδιαγραφές. Η τεχνική δυνατότητα δεν είναι πάντα εκείνη της μεγαλύτερης υποδομής και της μεγαλύτερης δυνατότητες παροχής. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το πώς μπορούν να αξιοποιούνται οι φυστάμενες εγκαταστάσεις και ε, τι γίνεται σε περίπτωση που σταματάει η ροή. Δεν μπορούμε να προσανατολιζόμαστε λοιπόν από τις μεγαλύτερες υποδομές, αλλά από τις κρίσιμες υποδομές, να βρούμε κάποια ευρυδική μορφή και φόρμουλα. Το ίδιο ισχύει και για την αλληλεγγύη. Ε, συνδέεται αυτό με τις περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί ε, αλληλεγγύη στην αγορά γενικώ, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τις λεπτομέρειες επιτόπου. Για να λειτουργήσει η αλληλεγγύη θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα κράτη να έχουν τον ίδιο ορισμό για τους προστατευόμενους πολίτες και τον ίδιο ορισμό για στάνταρ ε, εφοδιασμού. Τα είπατε και εσείς ο ίδιος. Η σημερινή πρόταση δημιουργεί μια θέση όπου καλούνται τα κράτη-μέλη να χαρακτηρίσουν όσο γίνεται περισσότερους πελάτες ε, προστατευμένους ε, για να μειωθεί η αλληλεγγύη. Και το άρθρο 12.2 ε, προβλέπει και κάποιο είδος απαλωτρίωσης. Και πότε μπορεί ένα κράτος μέλος να ε, προσφύγει ή να επικαλυστεί την αλληλεγγύη είναι έσχατη διαφυγή όταν θα έχουν χρησιμοποιηθεί και αποδεδειγμένα όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Όλα αυτά οδηγούν σε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, δεν ε, είναι σκόπιμα, δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν και να λειτουργήσουν. Το ίδιο ισχύει για την αλληλεγγύη μεταξύ γειτόνων. Σας το είπα και προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από το περιφερειακό στοιχείο και η άμεση γειτονία σου. Και μια τελευταία παρατήρηση για τη ροή. Βλέπω μια πρόταση που ε, είναι προσανατολισμένη πάρα πολύ στην υποδομή ή στις υποδομές. Αυτά όλα είναι αντιφατικά, βαριά στην εφαρμογή τους και γραφειοκρατικά. Ε, κατά θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, που έτσι και αλλιώς είναι αυτόματες για τη μεταφορά φυσικού αερίου, γιατί εκείνες... Ε, θα πρέπει να δώσουν ε, την έγκριση για το διαχειριστή τη λειτουργία του δικτύου TSO ε, σύμφωνα με την ε, νομοθεσία 2009 73. Δηλαδή, έχουμε πάρει εδώ μια βαριά για να σκοτώσουμε μια μίγα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια αναλογικότητα. Υπάρχουν και χώρες που δεν ειναι κράτη-μέλη της Ένωσης όπως η Ουκρανία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ και η κυρία Βέρνερ. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το 2006 και το 2009 που γνωρίσαμε ενεργειακές κρίσει, ε, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλε πρόοδοι στην ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου. Και οι δοκιμέ αντοχή στα stress test έδειξαν ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνα του να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ό,τι μέτρα και να λαμβάνουν. Καλωσορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω όμω να ε, επιμείνω σε τρία σημεία. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την κατανομή των κρατών μελών σε περιφέρειε. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπής ανεπιφύλακτα και επί της αρχής. Ε, και σε σχέση με τη δημιουργία μιας ε, κοινή ενεργειακής ένωσης είναι σωστό και χρήσιμο να ξεφύγουμε από την εθνική προσέγγιση και να περάσουμε σε μια περιφερειακή. Αυτό έχει συμβεί ήδη στον ηλεκτρισμό και σε σχέση με αυτά που είπε ο Κλοντ Τούρμες, ε, σε σχέση με αυτά που λέω συμφωνεί και η κυβέρνηση της χώρας μου. Και στην περιφερική κατανομή θα πρέπει να υπάρχουν και σχέδια ε, πρόληψης και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με τους γείτονες. Γιατί δεν είναι πάντα συμβατά τα συστήματα. Δεύτερον, Σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν μόνα του ποιου ε, πελάτε χαρακτηρίζουν προστατευόμενου. Το είπαν επανειλημμένα και προλαλήσαντε συνάδελφοι. Και εγώ θέλω μια ε, ε, ισχυρή εναρμόνιση θα πρέπει να είναι οι ίδιοι προστατευόμενοι πελάτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα χαιρόμουν το Κοινοβούλιο να προτείνει έναν νέο ορισμό. Για ένα τελευταίο και σύντομα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι χρειάζεται διαφάνεια στην υπογραφή συμφωνιών και συμβάσεων. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό πώς εξασφαλίζει ή βελτιώνει τον εφοδιασμό για την προμήθεια. Είναι γνωστό ποιε χώρε εξαρτώνται σε ποιο βαθμό από μεμονωμένου προμηθευτέ. Τι, τι δουλειά έχει διαφάνεια στα συμβόλαια, μπορεί να μα πει κάτι σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Κάριτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σε καλά χέρια η γνωμότηση αυτή, στα δικά σας δηλαδή. Έχοντας ακούσει και τους συναδέλφους Νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι στο φυσικό αέριο όπως γενικώ στην ενέργεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως νομοθέτες ώστε το κόστος ενέργειας να είναι όσο δυνατόν χαμηλότερο και για τη βιομηχανία και για τους πολίτες και να διατηρούμε την ανταγωνιστικότητά μας. Γιατί είμαστε σε μια παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει η ενεργειακή αγορά να λειτουργεί η αγορά του φυσικού αερίου να λειτουργεί και σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο. Και από αυτά που βλέπουμε από την ηλεκτρική ενέργεια, η περιφερειακή συνεργασία και οι περιφερειακές αγορές είναι κάτι πολύ σημαντικό και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι στο φυσικό αέριο εισάγουμε σχεδόν το σύνολο της κατανάλωσής μας. Μερικές από τις χώρες είναι σημαντικοί παίκτες στις αγορές, άλλοι, άλλες όχι. Η Ρωσία μέσω της Gazprom είναι πολύ σημαντική, η Νορβηγία επίσης. Και από αυτά που γνωρίζουμε από τις διακυβερνητικές συμφωνίες που εξέτασε η Κομισιόν, έχουμε πολλές παραβιάσεις και μιλούμε για διατάξεις ε, αντιμονοπολιακές. Ε, αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι αν θέλουμε μια ολοκληρωμένη αγορά φυσικού αερίου πρέπει να έχουμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να προστατεύουμε την αγορά αυτή. Και επομένω μιλούμε και για μεγάλες κλίμακος συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων. Όταν μια μεγάλη επιχείρηση που έχει 40% του μεριδίου της αγοράς προχωρεί σε μια συμφωνία, η Κομισιόν κάνει εξ ανάλυση. Εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε για εξάντε ανάλυση επί, στην περίπτωση τέτοιων συμφωνιών, τέτοιων συμβάσεων. Αυτές οι συμβάσεις συνάδουν με την ομοθεσία μας, διότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα, είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι όλα αυτά συνάδουν την νομοθεσία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ με τον κανονισμό αυτό κινούμαστε πιο κοντά στην Ενεργειακή Ένωση με ένα συντονισμένο σύστημα ασφάλειας εφοδιασμού αλλά βεβαίως είναι τμήμα μιας ευρύτερης δέσμης. Και έχουμε και την εμπειρία του προηγούμενου κανονισμού του 2010. Έχουμε λόγους να είμαστε πιο φιλόδοξοι, έχουμε τα αποτελέσματα των stress test, έχουμε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και διαμάχη στην Ουκρανία, έχουμε την προστασία των προστατευμένων καταναλωτών, την ε, αρχή της αλληλεγγύης δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εκεί πολύ ευέλικτοι σχετικά με αυτό. Αν πηγαίνουμε πολύ πιο πέρα από τα νοικοκυριά και πάμε και στις κοινωνικές υπηρεσίες, τότε το σύστημα εκτάκτου ανάγκης δεν θα είναι αποτελεσματικό. Και για τι αποζημιώσει και που είπε και ο κ. τηλίτσκα. Εδώ χρειαζόμαστε προληπτική δράση. Να, να εξασφαλίζουμε την αντίστροφη ροή, να έχουμε διαφάνεια, και να καλύπτουμε και μέρη της Ενιακής Ένωσης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τα κράτη να προχωρήσουν εθελοντικά σε ομαδοποιήσεις εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνολικά, ε, συμφωνώ με τη νέα πρόταση κανονισμού για νέα μέτρα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού του φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο ενωσιακό, προβλέποντας μηχανισμούς που θα μας προ... επιτρέπουν συντονισμένα να αντιμετωπίζουμε τυχόν διακοπές της ροής του εφοδιασμού. Και αυτό που, που προτείνουμε ως ε, πρώτη αντιμετώπιση της κατάστασης με την Ουκρανία και τη Ρωσία θα χρειαστούν ενίσχυση και βελτίωση. Επομένως, σύμφωνοι προς την ε, αρχή της αλληλεγγύης, οι έκτακτες ανάγκες θα πρέπει να εξασφαλίζουν φυσικό αέριο σε όλους τους ευάλωτους καταναλωτές και σε όλες τις ουσιώδεις υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Επί των προστατευμένων καταναλωτών, να διαφημίσω ότι στον ορισμό της κατηγορίας αυτής είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν και οι βιομηχανικοί τομείς για τους οποίους τυχόν διακοπή της ροής θα έφυγαν κινδύνο όλη, όλο τον κύκλο παραγωγής με δραματικές επιπτώσεις επί της απασχόλησης. Επίσης και πολύ σωστή η διάταξη η περιφερειακή. Εδώ χρειαζόμαστε συντονισμό ώστε να αποφύγουμε εθνικές επιλογές για την ασφάλεια του εφοδιασμού να έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί των γειτονικών χωρών. Και συμφωνώ με όσα είπε και η κυρία Γκρίφιν για τον Nord Stream. Συμφωνώ του με τα σχόλιά τη, Δεν θα τα επαναλάβω. Και υπογραμμίζω επιπλέον τη σημασία της οικοδόμησης μιας ολοκληρωμένης αγοράς για το υγρό φυσικό αέριο που είναι εναλλακτική δυνατότητα στους αγωγούς. Και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ενσωματώσει την πρόταση της Κομισιόν, αλλά εξασφαλίζοντας και την απαραίτητη συνάφεια με την ε, ενεργειακή ασφάλεια ώστε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε την εισαγωγή ορειτών καυσίμων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό κείμενο Είστε πραγματικός ε, ειδήμων σε αυτά τα ζητήματα, επομένω ε, δεν με εκπλήσει η ποιότητα της πρότασής σας. Όταν μιλούμε για την ασφάλεια εφοδιασμού, η αλήθεια είναι ότι εξετάζουμε παράλληλα πολλά ζητήματα. Η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού βεβαίως, ε, το ζήτημα της ελληνικής, αλλά και όπως είπαν ορισμένοι, είναι και τα όσα κάνουμε για την ενεργειακή απόδοση που είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση τομικών εφοδιασμού. Βεβαίω και υπάρχουν δίκτυα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ε, αγωγούς ε, και υποδομές. Σε ό,τι αφορά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Αυτό ο μηχανισμός αλληλεγγύη σε περίπτωση κρίση, όντω θα πρέπει να τον εξετάσουμε σε περιφερειακό επίπεδο, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, Όμω θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ορισμένα προσκόμματα. Για παράδειγμα, πώς ένας διανομέας μπορεί να εκτάσει παράλληλα μία ε, υποχρέωση αλληλεγγύη προ μια γειτονική χώρα και ταυτόχρονα ε, την προμήθεια ε, φυσικού αερίου στου ε, καταναλωτέ. Αυτό α πούμε είναι μια ιδιαίτερη διάσταση. Η περιφερειακή προσέγγιση είναι ενδιαφέρουσα λοιπόν, όμω θα μπορούσε να επιφέρει και έναν καταγερματισμό των αγορών. Όντω θα πρέπει να υπάρξει περιφερειακή προσέγγιση, αλλά να εξετάσουμε και μια ανώτερη προσέγγιση για ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Τέλος, να πω ότι ποτέ δεν κατακτούμε στο έπακρον την αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει συμπληρωματικά να έχουμε και τη συνεργασία με τους ε, σημερινούς προμηθευτές από τις επιμέρους τρίτες χώρες, αλλά ε, να βρούμε και νέους παρόχους από τη Μεσανατολή, την Κεντρική Ασία και το καθεξής. Επομένω, ε, πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί συνοχή σε διεθνέ επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ρόελ. Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, να πω μια άλλη σκέψη εγώ που μπορεί να έχει τη σημασία της. Αν δούμε σήμερα τον ε, εφοδιασμό σε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει αλλάξει σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε όταν αρχίζαμε τη συζήτηση ε, πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα δεν έχουμε έλλειψη αερίου και στο North Stream ρωτάμε αν χρειαζόμαστε όλη αυτή τη χωρητικότητα. Μήπως χρειάζεται, δεν χρειάζεται αυτό το έργο. Έχουμε LNG για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχουμε δυνατότητες προμήθειας παγκοσμίω, έχουμε διάφορους ε, προμηθευτές. Δεν είναι μόνο η Ρωσία που είναι το 30% ε, υπάρχουν και άλλοι, έχουμε και διαφοροποίηση. Λοιπόν, μήπως τώρα ε, το σημαντικότερο ερώτημα, πριν συζητήσουμε τα υπόλοιπα και την αλληλεγγύη και την κατανομή, το εξή ερώτημα. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη χωρητικότητα στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη από το τρίτο ενεργειακό πακέτο ή από υφιστάμενες οδηγίες και κανονισμούς αξιοποιούν όσο μπορούν την κατάσταση. Δεν έχουν μεταφερθεί παντού ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν κάνει αυτή τη δουλειά ακόμα. Ε, από εκεί θα άρχιζα εγώ. Και τουλάχιστον σε αυτό το κανονισμό θα το ανέφερα ότι το είναι ένα τώρα καθήκον είναι να ολοκληρώσουμε ε, τα όσα έχουμε ήδη νομοθετήσει. Εγώ δεν υποτιμώ τίποτα, αλλά λέω ότι ε, ε, κάθε πράγμα στο καιρό του και πρώτα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα και μετά το δεύτερο. Έχουμε και την αντίστροφη ροή και μια σειρά άλλες εξασφαλίσεις. Δεύτερον, εγώ είμαι υπέρμαχο αυτή τη περιφερειακής προσέγγιση. Πραγματικά είναι πολλά τα σωστά εδώ, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε τώρα ποιον θα παντρέψουμε με ποιον. Αυτό είναι το σημαντικό κριτήριο. Υπάρχουν ε, επιχειρήματα που συνηγορούν και προς τι δύο κατευθύνσει. Διασπορά κινδύνου. Επίσης σημαντικό επιχείρημα και θα πρέπει να το σκεφτούμε όταν συνενώνουμε χώρες. Ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Έχω πρόβλημα με ένα τρίτο σημείο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ποιε και πώ. Κοιτάξτε, είναι ιδιωτικέ αυτέ οι εταιρείε. Η Ευρώπη δεν είναι κρατική οικονομία, ούτε έχει τέτοια πρόθεση. Παλιά ήταν αυτά, περάσανε. Ε, ε, αν εποντάρουμε στην ιδιωτική οικονομία, τότε το θέμα είναι ποιο διαπραγματεύεται με ποιον, ποιο αγοράζει πώ και ποιο υπογράφει συμβάσει. Προσοχή. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επίγουσες καταστάσεις, αλλά δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε αποφάσεις για ε, ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα και τα και κοινέ προμήθειες με υπερβολική ενέργεια και πλεονάσματα. Εγώ διαφωνώ εδώ σε σχέση με μερικά που υπόθηκαν. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Μίστερ Κοχλίτσεκ νεοεκλεγής αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Έχω και εγώ μερικές παρατηρήσεις να κάνω. Έχω μεγάλη πείρα στη βιομηχανία και καμιά φορά ακούω διάφορα πράγματα που με κάνουν αμυδιό. Μετά την κρίση που γνωρίσαμε στο φυσικό αέριο ε, ήρθε αυτή η πρόταση για το συγκεκριμένο νομοθετικό πακέτο για τη δικτύωση ε, των κρατών των υποδομών. Έγινε αυτό. Μετά έγινε η νομοθεσία για την αποθήκευση φυσικού αερίου για ένα τρίμηνο. Όταν τα κράτη-μέλη δεν τα πληρούν αυτά, πώς να περιμένει κανείς αλληλεγγύη από τα κράτη αυτά. Γιατί εκτοτε έχουν παρέλθει έξι ολόκληρα έτη. Και ε, επίσης η αντίστροφη ροή θα πρέπει να ισχύει για όλα τα τμήματα του συστήματος. Ε, ε, και οι υποδομές φυσικού αερίου είναι θέμα των κρατών και των μεγάλων εταιριών. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε μια χώρα να αγοράσει φυσικό αέριο από μια άλλη χώρα από την άλλη άκρη του κόσμου. Αυτά είναι ανέκδοτα. Ε, αλληλεγγύη είναι, αλλά συμμετέχουν όλοι στην αλληλεγγύη. Όταν κάποιοι δεν εφαρμόζουν ε, τις συμφωνίες, έρχονται και μας ζητούν στη συνέχεια να κάνουμε ειδικέ ρυθμίσει για ειδικέ χώρε όπω είναι η Ουκρανία. Ή σου λένε ότι ο δεύτερο αγός Nord Stream είναι περιττός. Αφήστε να το αποφασίσουν αυτό εκείνοι που επενδύουν. Εμά τι μα νοιάζει, τι λόγο μα πέφτει. υπάρχει και αλληλεγγύη ανόητη. Ας πούμε, στην ε, ηλεκτροδότηση ε, ε, υψηλής τάσεως ε, πώς επιβαρύνεται ιδιαίτερα το δίκτυο στη Γερμανία από την νότια προς τη βόρεια Γερμανία. Στην Τσαχία είναι αλλιώ τα πράγματα με μετασχηματιστές και με άλλο τρόπο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, πριν αποφασίσουμε και βγάζουμε και διάφορα πορίσματα, θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Ε, είμαστε η οικονομία της αγοράς, δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Ε, καλή ενεργειακή ένωση, αλλά ε, είναι προβληματική η προμήθεια στην ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέβαν Μόζαρ, ε, στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας για τα ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού ενέργειας. Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ για την ευκαιρία που μας δίνετε να εξετάσουμε τον κανονισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού και σας ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια αυτή συζήτηση για το τι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Από δική μας σκοπιά αναγνωρίζουμε απολύτως ε, τη σημασία καλύτερης εφαρμογής ε, της, ε, πρώτης, της δέσμης μάλλον για την ε, ενεργειακή ασφάλεια και εξετάζουμε την ασφάλεια φοδιασμού σε ευρύτερο πλαίσιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο στην ενεργειακή απόδοση, στους κλιματικούς μας στόχους, στους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά αυτή φέτος ε, για να κάνει περισσότερες προτάσεις ακριβώς για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες και στο πλαίσιο της, πακε... μέτρων ε, για τον ε, σχεδιασμό της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε την ενεργειακή απόδοση ως κύριο μέσο για την επίτευξη της καλύτερης ασφάλειας εφοδιασμού. Είναι λοιπόν μια πρόκληση να δούμε πώς μπορούμε να κατανείμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, το φυσικό αέριο που έχουμε και που χρειαζόμαστε. Βασικό επίδευμα κατά τη γνώμη μας ενός βελτιωμένου κανονισμού θα ήταν η βελτιωμένη περιφερειακή συνεργασία. Ούτως ώστε τα κράτη-μέλη εκείνα που είναι αρκετά δυνατά να συνεργαστούν με εκείνα που έχουν αδυναμίες, ας πούμε που ε, παρουσιάζουν πλήρη εξάρτηση από έναν ε, προμηθευτή. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Να δούμε πού μπορούμε να πετύχουμε την ε, μεγαλύτερη προσθεμένη αξία και να διατηρήσουμε φυστάμενες πρακτικές σε άλλα κρατημέλη όπου ήδη υπάρχει κάποιο είδη συνεργασία. Επομένω, δεν θέλουμε να τα υποκαταστήσουμε όλα αυτά, αλλά να τα συμπληρώσουμε με άλλες ε, δυνατότητες για να σημειωθεί καλύτερη δυνατή πρόοδος ως προς ε, το σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο και εμείς αναγνωρίζουμε τι προκλήσει που αναφέρατε κι εσεί ότι οι περιφέρειες μπορούν ε, να ε, δημιουργήσουν κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε όλα αυτά με αρμονικό τρόπο να εντάσσονται στην ενεργική αγορά. Γι' αυτό έχουμε και εκθέσει αξιολόγηση ομοτήμων από εξωτερικού φορεί και θέλουμε να δούμε πώ ακριβώ θα προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά και να δούμε αν θα προκύψουν τυχόν προβλήματα από τα μέτρα που θα υιοθετηθούν στην περιφέρεια ε, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά άλλες περιφέρειες. Και θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη διαβούλευση διασυνοριακά κατά τη θέσπιση των μέτρων όταν θα προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα και μετά όταν θα ε, προσδιορίζονται και τα περιφερειακά μέτρα. Επομένω, θα πρέπει να το εξετάζουμε και διασυνοριακά αλλά και διαπεριφερειακά. Ε, για τους προστατευόμενου καταναλωτές και πελάτες, αναγνωρίζουμε τα όσα αναφέρετε, τι επιφυλάξει σα για ε, το βαθμό εναρμόνιση που απαιτείται. Έχουμε λάβει μια ενδιάμεση προσέγγιση Έχουμε εντοπίσει ορισμένα κρίσιμα σημεία, αλλά αφήνουμε και να περιθώριο ευελεξή τα κράτη-μέλη, γιατί ε, διαφέρει η κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την κατάλληλη ισορροπία. Γι' αυτό μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω να συζητήσουμε και μαζί σα και με τα κράτη-μέλη πώ μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Όμω δεν είμαστε πεπισμένοι ότι, ότι απαιτείται πλήρη συναρμόνιση. Η αλληλεγγύη σημαντική βελτίωση της πρότασής μας κατά τη γνώμη μας, εάν υιοθετηθεί, ως ε, απότερος μηχανισμός ε, διασφάλισης που βασίζεται σε πλήρως αρμονισμένα κριτήρια. Ε, προστατεύει μόνο τα νοικοκυριά και κανέναν άλλον. Δεν είναι το ίδιο με τους ε, προστατευόμενους πελάτες. Κύριο στοιχείο είναι ακριβώς η προστασία των νοικοκυριών, γιατί είναι η πλέον ευάλωτη... Ε, καταναλωτέ σε μια κρίση φυσικού αερίου. Επομένω, αυτοί θα πρέπει να προστατεύονται σε περίπτωση κρίσης και θα πρέπει ε, να βασιζόμαστε σε γειτονικούς ε, παρόχους της περιφέρειας. Με τα ενεργειακή κοινότητα που αναφέρθηκε και για μας είναι κέρια σημασία ζήτημα, να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και να λειτουργήσουμε και διασυνοριακά και να υπάρχει ε, καλή αμοιβαία συνεργασία. Και δίκαιη μεταχείριση των προμηθευτών. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την αποζημίωση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο των περιφερειακών σχεδίων. Και τα κάτι μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν ακριβώς ε, τους ε, συγκεκριμένους μηχανισμούς. Δεν έχουμε κάποια μαγική λύση αυτή τη στιγμή ε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, ο ανταγωνισμός πάντα ενέχει και ε, την τιμή της αγοράς και ένα, top up, ένα συμπληρωματικό ποσό ε, που θα χορηγείται κατά περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι φορά τη διαφάνεια των συμβάσεων, Είναι κάτι το οποίο εντάσσεται ε, ακριβώς στο ευρύτερο πλαίσιο, η βελτίωση των πληροφοριών. Θέλουμε να, όλες οι αποφάσεις να βασίζονται ε, σε μια πλήρη εικόνα με πληροφορίες ε, που προκύπτουν και από πτυχών ε, περιορισμούς που προκύπτουν από τις συμβάσεις. Δεν θέλουμε εμείς να πανεμβούμε βεβαίω στις ίδιες τις συμβάσεις, αλλά να εξετάσουμε τις συνέπειες ε, των συμβάσεων και να δούμε εάν μπορούμε να μετριάσουμε περιορισμούς ε, με άλλα μέτρα στο περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν πρόκειται για σύστημα κυρώσεων για τις συμβάσεις λοιπόν. Αυτό εναπόκειται στο δίκαιο ανταγωνισμού και ήδη φύσταται, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Τέλος, διαφοροποίηση. Κύριος πολιτικός στόχος. Εδώ και θεωρούμε ότι με αυτόν τον κανονισμό θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ε, για να κατανέμεται το φυσικό αέριο με αποτελεσματικό τρόπο και να έχουμε κατασκευή νέων υποδομών μόνο όπου αυτό είναι απόλυτο απαραίτητο, να αποφύγουμε την κατασπατάληση πόρων και να έχουμε καλύτερη ασφάλεια για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα κάποια λεπτά. Ο κύριος Σέριξον ήθελε κάτι να ρωτήσει. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο είχα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή για τον εφοδιασμό και την ασφάλεια του φυσικού αερίου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μιλούμε για το φυσικό αέριο ως λύση στο ευρύτερο κλιματικό ζήτημα και ως μετάβαση από το πετρέλαιο και το κάρβουνο, γιατί έχουμε μικρότερες εκπομπές, συχνά σκεπτόμαστε λίγο στενά και προς την λανθασμένη κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τις εκπομπές ε, αερίων στα κέντρα ενέργειας, στα εργοστάσια. Δεν είναι μόνο θέμα του Nord Stream. Μεταφέρεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα το φυσικό αέριο. και η υποδομή στη Ρωσία είναι πολύ παλιά με διαρροές παντού. Αν δείτε λοιπόν το σύνολο των εκπομπών όλου του συστήματος είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι στο επίπεδο των καταναλωτών ή των ε, μονάδων. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Να πω και εγώ δύο λόγια στο κλείσιμο της συζήτησης αυτής ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους 21 συγκεκριμένες παρατηρήσεις των σκιωδών μέτρησα και 12 ακόμα από τους υπόλοιπους. Πολλές λοιπόν παρατηρήσεις, πολλά σχόλια. Σας ευχαριστώ για μια θερμή συζήτηση. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εγώ είμαι απόλυτα προετοιμασμένος για αυτήν. Όπως ακριβώς το είπε η Τερέζα και έχει δίκαιο, είναι απολύτως σωστό ότι υπηρετούμε τους καταναλωτές, ναι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ε, επιχειρήσεις ενέργειας στην Ευρώπη. Ιδάλλως δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές. Η ισορροπία είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητη. Μιλούμε για την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της οικονομίας. Γιατί η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την ενέργεια, την ασφάλεια φαδιασμού, τις κατάλληλα συγκρατημένες τιμές, τη βιωσιμότητα. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική και χρειαζόμαστε και ασφάλεια και εναλλακτικές λύσεις εκτός από το φυσικό αέριο και για τις ανανεώσιμες πηγές. Θα μπορούσε να είναι ένα success story ευρωπαϊκό, όπως ήταν και ο πρώτος κανονισμός πριν από 6 χρόνια και είχαμε αμφιβολίες και πολλοί από εμάς θυμούνται και τις συζητήσεις τότε, δύσκολες συζητήσεις. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και ο κανονισμός εφαρμόστηκε. Και ακόμα περισσότερο από την τρίτη νεακή δέσμη το 2009, ακόμα νωρίτερα από τον κανονισμό μας του 10. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. 13 Ιουνίου είναι η επόμενη συζήτηση στην Ήτρε επί τη βάση του σχεδίου εκθέσεως ε, με όλες βεβαίως τις μεταβράσεις και προθεσμία για τις τροπολογίες δύο ημέρες αργότερα, 15 Ιουνίου. Εξέταση των τροπολογιών 11 Ιουλίου, ψηφοφορία στην Ήτρε τον Οκτώβριο έχουμε ένα πολύ αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Όπως και στην περίπτωση των 700 MHz του προηγούμενου θέματος. Τώρα λοιπόν είναι 11 η ώρα. Θέλετε μία φράση πριν το επόμενο θέμα. Δεν θα ήταν καλό για το θέμα αν έχουμε μία παρουσία έναν εκπρόσωπο της Ολλανδικής Προεδρίας. Το βλέπω λίγο, μου φαίνεται περίεργο ότι δεν είναι εδώ κανείς. Έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος και ενημέρωσα την Ολλανδική Προεδρία από την αρχή της ε, εντολής μας. Είχα συζητήσει εκπροσώπους, συζητήσαμε το φάκελο αυτό και συμφώνησαν ότι είναι πολύ σημαντικό και για εκείνους και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις συζητήσεις εξ όσων γνωρίζω από το Μάιο. Η Σλοβακική Προεδρία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου με την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα είναι σχεδόν από την αρχή του εξαμήνου. Ευχαριστώ. Ε, συναδελφοί, ευχαριστώ και ιδιαίτερα τους Σκιώδης για τη συνεργασία. Πάμε στο υπαριθμόν 5 ένας μηχανισμός ανταλλαγή ε, πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικέ ε, συμφωνίες και τα μη δεσμευτικά μέσα μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών ή στο πεδίο της ενέργειας με την κατάργηση της απόφασης 994 κάθετος 2012 κάθετος Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ε, Κρασνοντέψκι είναι εισηγητής και μαζί με τον προηγούμενο φάκελο εδώ βρισκόμαστε στο, στην ενεργειακή δέσμη, στη δέσμη ενεργειακής ασφάλειας μαζί με εκείνη φυσικού αερίου. Εδώ ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την, ε, την συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια των συμφωνιών αυτών διακυβερνητικών όπως και τη σχέση κόστος-οφέλους συνολικά και την ανταγωνιστικότητά μας. Ο πρώτος ομιλητής είναι βεβαίως ο ίδιος ο εισηγητής, ο κύριος Κρασνοτεύσκη. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος από ελληνικά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να πω δύο λόγια για αυτήν την ε, γνωμοδότηση που συντάσσω αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση της, ε, IADA, της απόφασης IADA είναι απαραίτητη για τη διάρκεια της ε, ανάλυσης αντικτύπου, IGA μάλλον, γιατί είδαμε ότι αυτή, σε αυτή τη φάση συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διακυβερνητικές συμφωνίες, αλλά δεν μας επιτρέπει να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα Υπάρχουν κάποιες στοιχεία των συμβάσεων αυτών δηλαδή που ενδεχομένως να μην συμμορφούνται προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά δυσκολευόμαστε να επιδιορθώσουμε την κατάσταση λόγω του περιορισμού που έχουμε στην αξιολόγηση των συμβάσεων αυτών και στην πρόταση του σχεδίου υπάρχουν κάποια ουσιώδη στοιχεία που θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μας πιστεύω γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες ως συνήθως και θα είναι το καθήκον του Κοινοβουλίου να εξετάσει αυτές τις δύσκολες λεπτομέρειες και ίσως να υποβάλει μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Θα μπορούσα όμως να υπογραμμίσω κάποια από τα πιο θετικά στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι η αξιολόγηση των IGA θα πρέπει να είναι εξάντε. Δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να αποφύγουμε κάποιες παγίδες. Παγίδες που θα μπορούσαν ε, να μας αποτρέψουν από το να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο, επίσης πολύ σημαντικό, είναι η πρόταση ότι όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τη σύμβαση αυτή, τη συμφωνία αυτή, θα πρέπει επίσης να αξιολογούνται. Δεν μιλούμε λοιπόν μόνο για την εκτίμηση της ίδιας της διακυβερνητικής συμφωνίας, στρίκτου sensu, αλλά και όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που τη συνοδεύουν, που επίσης θα πρέπει να αξιολογεί η Κομισιόν προκειμένου να καταλέξει το συμπέρασμα ότι συμμορφούνται προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εγώ το θεωρώ αυτό ουσιαστικότατη πτυχή. Ένα τρίτο στοιχείο που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αξιολόγηση των συμφωνιών αυτών ως προς την συμμόρφωσή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι η πρόταση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή και σε μη δεσμευτικά μέσα. Θα καλύπτονταν δηλαδή από τις συμφωνίες αυτές και μη δεσμευτικά μέσα. Αν έχουμε δηλαδή μια άλλη μορφή εκτός της IGA για τη συμφωνία, τότε η Κομισιόν προτείνει εκτός από την εξπόστ κοινοποίηση των εγγράφων αυτών, Θα μπορούσαμε ίσως να ήμασταν λίγο πιο φιλόδοξοι και εδώ. Θα μπορούσαμε δηλαδή να εξετάσουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των μη δεσμευτικών αυτών μέσων προκειμένου να αξιολογήσουμε τι θα μπορούσε να συμβεί, να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία θα κρίνονταν ότι δεν συνάδουν θα, θα κρινόταν ότι δεν συνάδουν αυτά τα μέσα προς τον ευρωπαϊκό δίκαιο, προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι θα συνέβαινε τότε. Συνοψίζοντας λοιπόν θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόταση συνολικά, μια απαραίτητη πρόταση, Και εδώ το κεντρικό σκεπτικό είναι να επιδιορθώσουμε, να καλύψουμε κάποια κενά και να εξασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές θα συνάδουν προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού των κρατών μελών. Συντοποιούμε βεβαίως όλοι ότι έχουμε κάποια προβλήματα υβριδικών συμφωνιών που δεν είναι πραγματικά εμπορικές συμφωνίες ή κρατικές διακυβερνητικέ και ίσως υπογράφονται σε παιδεία ή σε τομείς που δεν υπάρχονται σε έλεγχους. Και στην περίπτωση της ε, γνωμοδότησης του, του κυρίου Μπούζεκ είπαμε πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά για να τα ε, φέρουμε και εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο Πρόεδρος, για την παρουσίαση. Τώρα ο κύριος Μπουρούτσεφ από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι ε, ε, και πρόεδρε. ορίζω την νέα πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής προφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τα μη δεσμευτικά μέσα. διότι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Ιδιαίτερα την ασφάλεια εφοδιασμού και ε, ανταγωνιστικό κόστος. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό για να βγει καλός κανονισμός και χάρη στη συγκεκριμένη πρόταση να φτάσουμε πιο κοντά στην επιθυμητή εσωτερική αγορά ενέργειας. Η πρώτη νομοθεσία σχετικά θεσπίστηκε το 2012 όταν συμφωνήθηκε να γίνει μια επισκόπηση και θεώρηση των εφισταμένων διακυβερνητικών συμφωνιών. Είχε νόημα τότε και σημασία να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες και να εντοπιστούν τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την ασυμβατότητα ε, και τη μη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο. Η εκ των όμως κοινοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκεί πλέον σήμερα, γιατί έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Στόχο είναι η ολοκληρώση τη Ενεργειακή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν οι κοινοποίησει να έρχονται εκ των προτέρων ε, για τι κυβερνητικέ συμφωνίε ενώ και όχι απλώ ανακοίνωση αυτή τη στιγμή έχει συναυθεί μια συμφωνία. Τώρα στο Συμβούλιο γίνεται μια συζήτηση για τα, και για τα μη δεσμευτικά μέτρα. Ε, ε, τα κράτη-μέλη έχουν συμφέρον, πιστεύω, να έχουν ε, την ε, πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραστάτη στο πλευρό τους για να δούμε ε, ποιες είναι αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες και όταν διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες να το τσεκάρουν αυτό κατά πόσο είναι σύνομο με το ενωσιακό δίκαιο. Επαναλαμβάνω εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων, γιατί μετά είναι κατόπιν εορτής. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να εξασφαλίσει ε, καλύτερο ενεργειακό εφοδιασμό και πιο ασφαλή σε τιμές ανταγωνιστικές και προσιτές και να προστατεύει μια εσωτερική ενιαία ενεργειακή αγορά που να λειτουργεί απρόσκοπτα. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εκ των προτέρων προσέγγιση και όχι εκ των υστέρων και χαίρομαι για τους συναδέλφους που ξέρω ότι θα βοηθήσουν να καταληξούμε σε μια πολύ δυνατή και στεναρή στάση. Ευχαριστώ και θέση. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επίσης και ο δεσηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο εφιστάμενος μηχανισμός ε, με βάση τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις συμφωνίες μετά την υπογραφή τους ε, δεν λειτουργεί καλά γιατί δεν ε, διασφαλίζεται ότι αυτές οι συμφωνίες συνάδουν και συμφωνούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Συγητή και συζητήσαμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ε, δυνητική ή υποχρεωτική ρήτρα, may or shall. Και ε, αρχικά είχαμε επιλέξει το shall. Τώρα μετά από τέσσερα χρόνια εμπειριών καταλήγουμε στο ίδιο ερώτημα. Πώς θα πρέπει να αξιολογούμε τις διακυβερνητικές συμφωνίες. Και έτσι χαιρετίζω τις προτάσεις ε, του εισηγητή για τα όσα θα πρέπει να τροποποιηθούν. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί ορισμένα κρατημέλη έχουν δικές τους προτεραιότητες και ορισμένες φορές τα κρατη ενδέχεται να μην γνωρίζουν ε, τι όρους ε, επιτυγχάνουν κρατημέλη από τρίτες χώρες. Το έχουμε δει και εμείς, ότι έχουν υπάρξει περίεργες ε, συμφωνίες μεταξύ επιμέρους κρατών μελών και έχουμε άλλες προϋποθέσεις να ισχύουν για, τα, για τις χώρες της Βαλτικής και άλλες, ε, ε, με άλλους όρους να υπογράφουν μεγαλύτερα κρατημέλη. Ανέφερε η την ανάγκη συμπερίληψης μη, δεσμε, δεσμευτικών μέτρων στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που επιτρέπει ε, την παράκαμψη του ευρωπαϊκού δικαίου. Να κλείσουμε δηλαδή αυτά τα παραθυράκια και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κλείσουν. Ελπίζω να επιληθεί αυτό το ζήτημα άπαξ και διαπαντός. Και αυτό θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε πραγματική ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αμλίνερ Εσκιώδης, ε, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε σήμερα για αυτό το ζήτημα. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι προκειμένου να διαμορφώσουμε μια συμπεριληπτική ενεργειακή ένωση και να διασφαλίσουμε την ε, ενεργειακή ασφάλεια για του Ευρωπαίου πολίτε, θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαφάνεια των ε, ενεργειακών ε, συμφωνιών και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό προβλέπεται και από τον υφιστάμενο μηχανισμό. Όμω, ε, απεδείχθη ανεπαρκής για να επιλύσει το ζήτημα τη έλλειψης συμμόρφωσης των ενεργειακών συμφωνιών με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το κύριο πρόβλημα ήταν η καθυστερημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο πλαίσιο μιας εξπόστε αξιολόγηση των συμφωνιών. Για να επιληθεί αυτό το ζήτημα, η υποχρέωση υποβολή εκθέσεων για τις συμφωνίες θα πρέπει ε, να βελτιωθεί. Ένας απλός μηχανισμός ε, ενημέρωση δεν θα οδηγήσει σε συμμόρφωση εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ενημερώνεται για τη συμφωνία πριν την κύρωσή τη. Γι' αυτό θεωρώ ότι μία ε, πιο έγκαιρη ε, συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία θα ήταν χρήσιμη, γιατί έτσι θα ενισχύσουμε και τη διαπραγματευτική ισχύ των κρατών μελών. Ε, υπάρχει ανάγκη καλύτερη εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την εξάρτηση από ενεργειακού παρόχου. Όμω θα πρέπει να βρούμε και μια ισορροπία και μια λογική προσέγγιση που θα προστατεύει τα κράτη-μέλη από την υπογραφή μη ευνοϊκών συμφωνιών με τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα θα σεβόμαστε πλήρως και το δικαίωμα των κρατών μελών να συνάπτουν μεμονωμένες ε, συμφωνίες. Έτσι θα αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και θα έχουμε και πιο φτηνή ενέργεια για τους Ευρωπαίους πελάτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τούρμες εκπροσωπώντας του πρασίνους ως κοιότης. Ευχαριστώ. Εξ του κυρίου Ταράντ παίρνω τον λόγο που θα διαπραγματευτεί το φάκελο ε, από πλευράς ομάδας μας. Ο Nord Stream και όλες αυτές τις συζητήσεις δείχνουν ότι τέτοιου είδου ε, συμβάσεις είναι κάτι παραπάνω από εμπορικές. Δεν μπορούμε ε, να αποκρύψουμε αυτόν τον διαφορετικό χαρακτήρα και να λέμε ότι είναι μόνο πολιτικές συμβάσεις, γιατί έχουν και γεωπολιτικές επιπτώσεις και το βλέπουμε και από το Nord Stream και όλες τις ε, επιπτώσεις που έχει για την Ουκρανία ε, και το πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη. Είναι ενδιαφέρον. Τελευταία φορά χάσαμε το Shell εξαιτίας της Shell. Δηλαδή οι ίδιες εταιρείε είναι αυτές που μας αποτρέπουν να κάνουμε μια καλή συμφωνία. Τώρα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση και χρειαζόμαστε αυτή την εξάντια αξιολόγηση. Είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε όχι μια φωνή. Χρειαζόμαστε 29 που θα όμως αποστέλουν ένα κοινό μήνυμα και θα διπραγματεύονται από κοινού. Και αυτό γίνεται μόνο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργήσει ως συντονιστής. Και στην Πολωνία είχαμε μια πολύ καλή εμπειρία στην τελευταία τέτοια διαπραγμάτευση. Και αν δείτε πόσο καλύτερη έγινε η συμφωνία τελικά, γιατί ε, μιλήσαμε με την ε, σορευμένη ισχύ της Ευρώπης και όχι μόνο μία χώρα ε, έναντι της Ρωσίας. Αυτή λοιπόν είναι η λύση και μία θετική ε, επίπτωση αυτής της επιλογής. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ευρεία οτι θα υπαρξει μια ευρία πλειοψηφια στο Κοινοβούλιο για να επιψηφιστεί. Είμαστε ε, μαζί με την Επιτροπή και θα υπάρξει και καλή πλειοψηφία πιστεύω στο Συμβούλιο. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία για τη νέα πολωνική κυβέρνηση για να δει ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια και να το ανήκει κανείς ε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι κάτι το θετικό και υποφελές. Και Τζέρσι, όταν οριστικοποιήσουμε την ε, ε, συμφωνία μπορούμε να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Σημαία στη Βασοβία και ίσως να μας επιτρέψουν να βάλουμε στο Πολωνικό Υπουργείο Ενέργειας δίπλα-δίπλα την Ευρωπαϊκή και την Πολωνική Σημαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Σε ευχαριστώ για τη σχόλιά σου. Από πλευράς Γκουε, σκιώδης συζητητής, ο κύριος Λυκιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω ότι για την ομάδα μα, την ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, η πρόταση τη Κομισιόν για τι διακυβερνητικέ συμφωνίε περιλαμβάνει πολλέ αρνητικέ αναφορέ. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα για μα είναι προβληματική πρόταση να εμπλακεί η Κομισιόν στι διαδικασίε πριν από τη σύναψη συμφωνιών και να είναι υποχρεωτική η εκ των υστέρων αλλά και εκ των προτέρων αξιολόγηση των συμφωνιών από την Κομισιόν. Εμεί διαφωνούμε με την πρόταση τα κράτη-μέλη να είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν την Κομισιόν ακόμα και για την πρόθεσή του να αρχίσουν διαπραγματεύσει. Καθώ και με την πρόταση τα αιτήματα των κρατών μελών για ιδανό όσον αφορά συγκεκριμένε πληροφορίε να μην περιορίζουν την πρόσβαση τη ίδια τη Κομισιόν σε αυτά. Οι εν λόγω προτάσει περιορίζουν την κυριαρχία των κρατών και υποβαθμίζουν τον ρόλο του καθώ πλέον θα υπάρχει πλήρη εξάρτηση από την Κομισιόν και καμιά ενέργεια δεν θα μπορεί να γίνει από τα κράτη-μέλη χωρί τη σύμφωνη γνώμη τη. Δεν γίνεται τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να υπογράφουν, να κυρώνουν, ούτε καν να συνομολογούν τα σχέδια των διακυβερνητικών συμφωνιών όπω ζητείτε στην πρόταση που έχει καταδεθεί. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση μια ενεργειακή πολιτική η οποία ελέγχεται από την Κομισιόν και να περιορίζει την εθνική ευελιξία στη διαμόρφωση πολυδιάστατων αποδοτικών διακρατικών ενεργειακών σχέσεων. Και ξέρετε γιατί. Ιδιαίτερα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε ακόμα να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην ενεργειακή τροφοδοσία σε πολλά κράτη και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα υπάρχουν κράτη, μέλη και περιοχές που είναι απομονωμένα από τα ενεργειακά δικτυά και παρόλα αυτά ζητείται να υπάρχει έλεγχος στις διακρατικές συμφωνίες. Ε, γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι αρνητικά. Θα μπορούσε να μιλούμε για αυτή τη διακρατική συμφωνία, αυτή την συνεννόηση και τον συντονισμό, εφόσον λύσουμε τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την απομόνωση και την ασφάλεια. Για μα είναι σημαντικό να ενισχύσει να υπάρχει πρώτα-πρώτα δημόσιο έλεγχο στα δίχτυα, στι συμφωνίε, τι διακρατικέ, να προωθούνται διεθνεί συνεργασίε στη βάση του αμοιβού ωφέλου και τη αλληλεγγύη και προ αυτήν την κατεύθυνση θα καταθέσουμε τι τροποποιήσει μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Oh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφα. Ο κύριος από ε, το EFTD, ο Σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο ανταλλαγής ε, για το θέμα αυτό, νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε και σε θέματα που θεωρούνται δευτερεύοντα ε, στο πλαίσιο της εργασίας της και μιλώ για την πρόταση διπλής υποχρέωσης που θα επιβάλλεται σε κράτη-μέλη. Καταρχάς, εξ αντεκοινοποίησης ενδεχόμενων ενεργειακών συμφωνιών με τρίτους εταίρους και τις ενδείξεις και τα υπόλοιπα έγγραφα που θέλει η Κομισιόν στα πλαίσια των ιδίων συμφωνιών. Εμείς εδώ περιμένουμε μια πολύ καλή δουλειά από τον εισηγητή σχετικά με τους μηχανισμούς και τις νομικές υποχρεώσεις. Και ιδιαίτερα λόγω του διαφοροποιημένου ειδικού βάρους ε, που δίνει και ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ. Αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε άλλες πτυχές της ε, ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σχετικά με τους ε, προστατευμένους πελάτες. Αν δεν είναι ερμονιστή αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε στρεβλώσεις εφαρμογής δικαιωμάτων και προστασίας της αγοράς χρειαζόμαστε να τηρούμε πάντοτε την αρχή της επικουρικότητας ώστε να λειτουργούν και οι περιφερειακοί φορείς αποτελεσματικά. Συμμεριζόμαστε λοιπόν το συνολικό στρατηγικό στόχο αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή και να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρόκειται για ένα στρατηγική σημασία θέμα που έχει αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας παντού, σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες λοιπόν και να μην απομακρυνόμαστε από τους συγκεκριμένους στόχους πολιτικής αυτής. Εδώ το θέμα δεν είναι μια πιο κεντρική διαχείριση, αλλά η καλύτερη προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τώρα συζητούμε την πρόταση αυτή και έχουμε ένα σοβαρό ε, πραγματικά ε, λίθο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που ε, έχουμε ένα κυρίαρχο προμηθευτή και δεν είναι εμπορική η παρουσία, αλλά είναι έντονα πολιτική στην προμήθεια της ενέργειας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει ένα μήνυμα. Δεν θα υπάρξει μάλλον δεν έχει υποβληθεί εθελοντικά ποτέ ένα σχέδιο κυβερνητικής συνεργασίας για έλεγχο εκ των προτέρων. Και αυτό και μόνο ε, συνιστά δικαιολογία και λόγο για υποχρεωτική κοινοποίηση εκ των προτέρων οποιασδήποτε διακυβερνητικής συμφωνίας. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και θα πρέπει να καλύπτει αυτό και τα μη δεσμευτικά μέσα, ε, όπως ε, λέγει η πρόταση. Εγώ είμαι υπέρ της ε, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις βεβαίως. Έχει δίκιο ο κύριος Τούρμελ, σε αυτό βοήθησε την Πολωνία στις δικές μας διαπραγματεύσεις και θα μπορούσε ενδεχομένω να βοηθήσει και τους άλλους. Ευχαριστώ. Thank you ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρινς. Είναι last minute αυτός ο μιλητής. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, υποστηρίζω αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία τη τελευταία φορά ήμουν εισηγητή όταν μιλήσαμε για τι διακυβερνητικέ συμφωνίε εκ των υστέρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και διαπίστωσε ότι το 1 τρίτο των διακυβερνητικών συμφωνιών αντιδίκεται στο κοινοτικό δίκαιο. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά και βαριά οι διαδικασίε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν συμφωνίε. Ε, Αυτή τη στιγμή έχουν υπογραφεί. Γι' αυτό λέμε να κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Γι' αυτό υπάρχει και ο ανταγωνισμό και το κοινοτικό, το ενωσιακό πλέον δίκαιο και θα πρέπει να τηρείται και να εφαρμόζεται. Εγώ έχω την υποψία ότι στο Συμβούλιο θα γίνει η καφγάς, όπως έγινε και την τελευταία φορά. Υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου και έχει απολύτως νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος, κανείς ζητεί το λόγο. Α, να παρακαλέσω τότε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το Διευθυντή, τη Γενική Διευθυνέργειας τι διευθύντρια, μάλλον την κυρία Μάχτιλτ Βέρστορφερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Κραστοντέσκη και όλου και όλε εισηγητές και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο. Όντω, οι διακυβερνητικέ συμφωνίε ε, πρέπει να συμμορφούνται πλήρως ε, με τις ε, διατάξεις και του ευρωπαϊκού δικαίου σε ό,τι αφορά την προμήθεια ενέργειας από τρίτες χώρες. Και το Μάρτιο και το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε φιλόδοξη πρόταση για πλήρη συμμόρφωση. Η πρόταση λοιπόν του 2012 για τις διακυβερνητικές συμφωνίες για την ενέργεια ε, ήταν πάρα πολύ στεναρή και από τον προηγούμενο εισηγητή όπως αναφέρθηκε για να έρθει εγκαίρος τον Οκτώβριο του 2012 μια καλή συμφωνία. Τώρα έχουμε αποκομίσει κάποια εμπειρία. 124 είναι αυτές οι συμφωνίες που έχουν κοινοποιηθεί και περίπου το 1 τρίτο χονδρικά δεν ήταν ε, ε, σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει οτιδήποτε εκ των υστέρων. Άρα, θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες, να κοινοποιούνται αλλά δεν αρκεί η εκ κοινοποίηση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Και λοιπόν προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Βασικές αλλαγές σε σχέση με το ισχύον σύστημα, πρώτη και σημαντικότερη, είναι να υπάρχει υποχρεωτική εκ των προτέρων ε, αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου διακυβερνητικών συμφωνιών και τα κράτη-μέλη θα απαγορεύεται να υπογράφουν ή να κυρώνουν σχέδιο τέτοια συμφωνία με τρίτη χώρα μέχρι να νομοδοτήσει η Ευρωπαϊκή χωρα μεχρι να αρμοδοτησει η ευρωπαικη επιτροπη για το κατά πόσο αυτό συμμορφούνται με το ενωσιακό δίκαιο και με τις ε, πολιτικές μας για την ασφάλεια ενεργειακό εφοδιασμό, για την ανταγωνιστικότητα και την νομοθεσία μας εν γέννη. Και επίσης εισάγουμε και μια υποχρέωση ε, να κοινοποιούνται εκ των υστέρων πια τα μη δεσμευτικά μέσα αυτό που δεν άλλαξε είναι ότι θα πρέπει ε, να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις. Όχι, δεν θα είναι. Για να μην στείλουμε λάθος μήνυμα στα κράτη-μέλη για τη συμβατότητα απριόρι. Δηλαδή, δεν προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις διαπραγματεύσεις στο πλευρό των κρατών μελών. Και επίση προτείνουμε να υπάρχει διαφάνεια στο σχετικό ε, ε, κανονισμό που συζητήσατε το πρωί και γενικά ε, πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ ισόρροπη η πρόταση. Να εξασφαλίζουμε ότι θα είναι σύνομε αυτέ αυτές συμφωνίε, συμφωνίες, πάντα σεβόμενοι την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν διεθνείς διακυβερνητικές διακρατικές συμφωνίες. Έχουμε ένα ευρύτερο πακέτο, μια δέσμη ε, για την εσωτερική αγορά ενέργειας, για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια στον εφοδιασμό. Είναι καλή συζήτηση, θα έρθει ε, στο Συμβούλιο. Ξέρετε ότι ε, στο Κοινοβούλιο, συγγνώμη, στο Συμβούλιο έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση στην ομάδα εργασία. Σήμερα ανταλλάσσετε εσείς απόψεις για πρώτη φορά, αλλά και το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου νομίζω θα μας επιτρέψει να γίνει γρήγορα η συζήτηση γιατί η πρόταση είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ. Κυρία Βέρσντορφερ για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Κρασνοντέψκη. Δεν ξέρω Έχετε να κάνετε καταληκτικά σχόλια, να προσθέσετε, να συνοψίσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, έχω καταγράψει όλα τα σχόλια και με χαρούπιν ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρθηκαν. Οι περισσότερε παρατηρήσει νομίζω τείνουν να συμφωνήσουμε με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πολύ θετικό. Βεβαίω υπάρχουν και διαφωνίε, αλλά με τα χαρά να τα εξετάσουμε από κοινού. Και μετά για τον εκπρόσωπο των Πρασίνων ήθελα να δώσω μια απάντηση. Έκανα ένα σχόλιο για την πολωνική κυβέρνηση και σε σχέση με την αλληλεγγύη και το καθεξής. Τέλος πάντων έφυγε, οπότε δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Έχουμε εξετάσει δι... τρεις εκθέσεις σήμερα το πρωί και οι τρει ήταν ε, στο... στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Επομένω, ε, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν στους επόμενους μήνες, όμως ε, στις 27 Ιουνίου του 2016 θα εξετάσουμε το προσχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Θα το συζητήσουμε λοιπόν περαιτέρω τότε και μετά θα εξετάσουμε και τις ε, τροπολογίες στις 5 Σεπτεμβρίου. Και 13 Οκτωβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε. Αυτό είναι το προσωρινό τουλάχιστον χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά αυτή τη έκθεση για τις διακυβερνητικές συμφωνίες και μη δεσμευτικά εργαλεία μεταξύ κρατών μελών και των χωρών στον τομέα της ε, ενέργειας και την ε, κατάργηση της απόφασης του 2012. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη μελέτη για την Ενεργειακή Ένωση κέρδιες αποφάσεις για την υλοποίηση μιας πλήρους ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας, παρουσίαση από τον κύριο Ράντε Μάκρης, και τον κύριο Νιούφελ. Έχουμε λοιπόν δύο εκπροσώπους της ε, εταιρείας Trinomics Consulting. Έχουμε λοιπόν τους δύο μιλητές που έχουν εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος ε, της Επιτροπής Ήτρε και των συντονιστών πιο συγκεκριμένα. Η μελέτη δίνει μια επισκόπηση και ανάλυση των βασικών ε, ευρωπαϊκών πολιτικών μέτρων και εργαλείων που συμβάλλουν ε, στην πλήρη ολοκλήρωση και εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Κρίσιμη σημασία λοιπόν για εμάς ε, μια τέτοια μελέτη και κάνει και ορισμένες ε, συστάσεις πολιτικής ε, για βελτιώσεις που μπορούμε να επιφέρουμε. Το έχουμε συζητήσει βέβαια και στο παρελθόν ε, αυτό το ζήτημα εκτενώς, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τους ομιλητές μας για να ακούσουμε και τις ε, δικές τους απόψεις για την ολοκλήρωση και εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και πιο συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία. Mm. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Κουν Ράντε Μάρκες ονομάζομαι, είμαι διευθυντής της Trinomics και έχουμε εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Αποκαινούμε μία ε, ισπανική συμβουλευτική, την Ήτρη, και ε, μία ουγγρική, την Energia Club. Ε, σκοπός της μελέτης ήταν, όπως βλέπετε και στις διαφάνειες, να εκτιμήσουμε σε ποιο βαθμό η... Ε, οι στόχοι για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μπορούν να επιτευθούν ε, με βάση τα υφιστάμενα μέτρα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι είναι η Ενεργειακή Ένωση και τι ρόλο διαδραματίζουν ε, οι επιμέρους πολιτικές και εργαλεία. Μπορείτε να τη βρείτε και σε έντυπη έκδοση στην είσοδο της αίθουσας. 60-70 σελίδες ε, είναι αυτή η μελέτη και σε αυτές τις σελίδες ε, περιγράφουμε σε εντομία το υπόβαθρο της Ενεργειακής Ένωσης ε, και τα όσα συμβαίνουν σήμερα και γιατί βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως ελπίζαμε ότι θα είναι πριν από μερικά χρόνια και έχουμε και ορισμένες συστάσεις. Στόχος λοιπόν είναι να περιγράψουμε το φάσμα των εργαλείων που διαθέτουμε, να εντοπίσουμε στενοπούς και να προτείνουμε συστάσεις για βελτίωση της πολιτικής. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι πολύ απλή. Βάσει ε, μιας συλλογής και ανάλυσης συναφών πληροφοριών και δεδομένων, ε, ε, νομοθετικά και κανονιστικά έγγραφα και ούτω καθεξής. Όμως, έχουμε συνεργαστεί και με εμπειρογνώμονες και στην Ανατολική και στην Νότια Ευρώπη Μιλήσαμε λοιπόν με πολλούς εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης. Έχουμε συνοδεύσει και συμπληρώσει ε, ως υπόβαθρο ε, και τρεις ε, μελέτες περιπτώσεων και studies. Αρχικά σε ό,τι αφορά την ε, σύζευξη των ε, των αγορών χονδρική στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναγκαιότητα και ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τους ε, μηχανισμούς ε, αποζημιώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και συνεργασία με την Acer και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτο case study, αντίκτυπος της ε, κατανομής χωρητικότητας εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ουγγαρία σε ό,τι αφορά την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είδαμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά πρέπει να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη ε, στην πράξη. Τώρα, σε μεγαλύτερο βάθος θα συνεχίσει ο συνάδελφος Λουκ Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα σταθώ σε ορισμένα βασικά ευρήματα και συστάσεις. Όπως παρατηρήσατε, έχουμε 11 βασικά πορίσματα και 11 συστάσεις στη μελέτη μας. Θα τις ε, παρουσιάσω βάσει τριών ομάδων. Πρώτα έχουμε τα δίκτυα ε, μετάδοσης ε, και διασύνδεσης και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να έχουμε μια ολοκληρω... για να έχουμε μάλλον μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας απαιτούνται ε, δίκτυα μετάδοσης και διασύνδεσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και γι' αυτό αποτελεί κύριο σημείο εστίασης της μελέτης μας. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή στόχος ε, για την ε, χωρητικότητα ε, διασύνδεσης. 10% λοιπόν της ικανότητας παραγωγής θα πρέπει να διατίθεται μεταξύ των μελών και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 8%. Επομένως, κατά μέσο όρο δεν έχουμε ακόμα πετύχει το στόχο που έχουμε θέσει το 2020. Και βάσει της μενής κατάστασης, Πολλοί φοβούμεθα ότι ο στόχος ε, του 2020 δεν θα επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα στόχο του 15% μέχρι το 2030, όμως εμείς ε, έχουμε κάνει ορισμένες παρατηρήσεις ε, για αυτό το στόχο. Προτείνουμε έναν ε, στόχο με γνώμονα ε, την οικονομική διάσταση που λαμβάνει υπόψη ε, και την παραγωγή, τις καμπύλες ζήτησης και τυχόν ωφέλη των σύγχρονων υποδομών διασύνδεσης. Για το φυσικό αέριο ξέρετε μάλλον δεν υπάρχει σαφή στόχος, όμως τα επίπεδα διασύνδεσης έχουν αυξηθεί ή αυξάνονται. χάρη στον κανονισμό ασφάλειας εφοδιασμού που προτείνει, ε, υποδομή, προβλέπει μάλλον υποδομή νήμιον 1 και οδηγεί σε σημαντικές υποδομές που αυξάνουν τα επίπεδα διασύνδεσης. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική προσέγγιση. Έχουμε τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ε, διασύνδεση των επιμέρους αγορών ε, και συστημάτων. Υπάρχει χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλά τέτοια μέσα. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εν γέννη ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση ε, παρέχει το 5% της απαιτούμενης χρηματοδότησης και των απαιτούμενων επενδύσεων. Σημαντική λοιπόν ε, συμβολή, αλλά το ευρύτερο πλαίσιο και επενδυτικό κλίμα μπορεί ακόμα να βελτιωθεί ε, για να προσελκύσει και ιδιωτικές επενδύσεις και για να διευκολύνει την ύπαρξη τέτοιων επενδύσεων. Σε αυτό το ε, πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί και η συνεργασία μεταξύ ε, των τοπικών αρχών. Η διασυνοριακή λοιπόν συνεργασία μεταξύ των επιμέρους διαχειριστών δικτύων μεταφοράς για να διευκολύνουμε και τις διασυνοριακές επενδύσεις, αλλά και για να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση και αξιολόγηση των οικονομικών ωφελών. Και το διοικητικό άκθος βεβαίως είναι ε, σημαντικό ζήτημα. Η δεύτερη κατηγορία. Συστάσεων και κύριων πορισμάτων ε, εστιάζεται στην ε, παραγωγή ενέργειας και την ασφάλεια εφοδιασμού. Βεβαίω, αν θέλουμε μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, απαιτείται ικανότητα παραγωγής. Και αυτό είναι κρίσιμο με αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι τα εθνικά ε, καθεστώτα στήριξη για τι ανάλογες πηγέ ενέργεια αφορούν και την επένδυση και στην συμβατική παραγωγή ενέργειας. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές αυτή τη στιγμή και οι, οι τιμές spot αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σήμερα είναι 24 με 26 ευρώ στο Βέλγιο, στο Μπέλπαξ και με μια τέτοια τιμή spot δεν μπορούμε να καλύψουμε και τις, ε, το μεταβλητό κόστος ε, της παραγωγής ενέργειας. Και δυστυχώ ούτε καν το πλήρε κόστο. Γι' αυτό, εν γέννη στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν πλέον επενδύσει στην συμβατική παραγωγή ενέργεια. Κάτι το οποίο όμω απαιτείται για να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού μέσω και μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή, στα περισσότερα κράτη-μέλη, ε, υπάρχει ικανή χωρητικότητα παραγωγής, παρότι στα προστακρατημέλη κράτη-μέλη είναι κρίσιμη κατάσταση. Σημαντικό θέμα σε αυτό το πλαίσιο είναι και το ίσο πεδίο ανταγωνισμού, απαραίτητο στοιχείο στο παρελθόν με τι μη απελευθερωμένε αγορέ και χωρί κανέναν ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών ενέργεια, αυτό δεν ήταν κρίσιμη σημασία θέμα. Σήμερα όμω υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμός στι περιφερειακέ αγορέ και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ίδιοι οι όροι ανταγωνισμού ω προ ε, την φορολόγηση τη ενέργεια ε, για την πρωτογενή ε, ενέργεια για παράδειγμα, αλλά και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των υποδομών. Και ξέρω ότι σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν φόροι στον άνθρακα, στο φυσικό αέριο, στην, υποδημές ε, παραγωγής ενέργειας, ακόμα και στην πυρηνική ενέργεια. Στη Σκανδιναβία υπάρχουν ακόμα ε, και φόροι για την ε, παραγωγή υδροληπτικής ενέργειας. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξουν επενδύσει, απαιτείται ένα σταθερό, προβλέψιμο και ευνοϊκό κλίμα επενδύσεων. Και αν ακόμα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, υπερεθνικό λοιπόν επίπεδο. Και ξέρετε ότι σήμερα κάποια κρατημέλη είτε εφαρμόζουν είτε εξετάζουν το δεχόμενο να εισαγάγουν έναν ε, μηχανισμό ανταμοιβή ω προ την ικανότητα, CRM. Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτό να υπάρχει ε, συντονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι εφικτό ή και πολιτικά αποδεκτό να έχουμε ενιαίο τέτοιο μηχανισμό CRM, όμως τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένα χαρακτηριστικά για να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο, πλαίσιο οποιοδήποτε τέτοιο μηχανισμό θα πρέπει να είναι ανοιχτός ε, για τη διασυνοριακή συμμετοχή, να αφορά ολόκληρη την αγορά, όλες τις τεχνολογίες, για να μην υπάρχει και στρέβλωση μεταξύ ε, εμπορευομένων και επιμέρους τεχνολογιών. Κλείνοντας, το πλέον ε, σημαντικό πλαίσιο παραγόντων είναι οι αγορές. Ξέρουμε ότι είναι ζήτημα ουσιαστικά κατάλληλη και σωστή ε, εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Έχουμε παρουσιάσει ένα case study ω προ ε, την ε, κατανομή ικανότητα εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ουγγαρία και εδώ είναι ένα από τα παραδείγματα όπου δεν τηρήθηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διατηρήθηκε η Εθνική Νομοθεσία για τέσσερα χρόνια, η οποία ε, δεν συμμορφώνεται με την ε, ευρωπαϊκή και αυτό ζημίωσε και την τοπική οικονομία και ούτω καθεξής. Και για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο υπάρχουν ε, πρότυπα με στόχους για την επιμέρους αγορές και αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν επιγόντως. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύσταση. Αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση των ε, αγορών χονδρικής βλέπουμε ότι ε, κινείται προς σωστή κατεύθυνση, υπάρχει πολύ σημαντική πρόοδος, όμως αυτή η πρόοδος καθυστερείται από την ανεπαρκή διακυβέρνηση, γιατί η υπερεθνική διακυβέρνηση είναι μάλλον αδύναμη. Έχουμε αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές, και ως συνέπεια της ε, αύξησης της χρήσης ε, και των ανανεώσιμων υπάρχει μεγαλύτερη συμφόρηση. Σήμερα λοιπόν ε, έχουμε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια και γι' αυτό απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις σε δίκτυα για να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση και να βελτιώσουμε την λειτουργία και την ολοκλήρωση των αγορών. Υπάρχουν λοιπόν ε, πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλευθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση, να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ αρχών και μεταξύ ε, των ε, διαχειριστών δικτύων και μπορούμε να συστήσουμε και την δημιουργία περιφερειακών TSOs τέτοιων διαχειριστών που να είναι αρμόδιοι ε, για την ε, διαδικασία κατανομής, για παράδειγμα. Τέλος, η τελευταία σύσταση αφορά τις αγορές λιανικής. Αυτό δεν συνδέεται βέβαια με την ολοκλήρωση ε, των αγορών, γιατί οι αγορές λιανικής είναι ακόμα εθνικές. Όμως έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά και απόκληση. Μόλις ένα τρίτο των αγορών λιανικής στην Ευρώπη μπορούν να θεωρηθούν ως δυναμικές. Ε, ένα τρίτο των αγορών ακόμα τη χάνουν Εντάξει, δεν είναι και μονοπόλια, αλλά δεν υπάρχει κανονικός συνταγωνισμός. Και ένας από τους ε, κύριους, ε, τις κύριες αιτίες έλλειψης ανταγωνισμού είναι ότι πολλές από τις ε, τιμές λιανικής ακόμα τη χάνουν ρύθμιση στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ ρύθμισης τιμών ε, και ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μηνύματα. Για να έχουμε ε, σωστές αγορές με εύρυθμη λειτουργία δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται οι τιμές. Και στις τιμές ενέργειας και στις υπηρεσίες ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να παρέχονται σε όρους που θα καθορίζονται από την αγορά. Συμπερασματικά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην λειτουργία και ολοκλήρωση των αγορών στην Ευρώπη, όμως πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, πολλά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ε, για να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, ομιλητές που παρουσίασαν τη μελέτη. Ας ξεκινήσουμε την συζήτηση. Κύριο Σκοβίτσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας. Μας μίλησε για δέσμευση χωρητικότητας και για την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, όταν παράγω εγώ μια ηλεκτρική ενέργεια όμως δεν μπορώ να την πουλήσω φθηνότερα στους άμεσους γειτονικού πελάτες σε σχέση με ε, κάποιους πιο μακρινούς πελάτες. Αυτό δεν έχει νόημα να παραδιδόμαστε στην αγορά. Όταν φτιάχνεις μια υποδομή φωτοβολταϊκά, ξέρω εγώ, ή μια ανεμογεννήτρια, δεν μπορείς να απαγορεύεις στους άμεσους γείτονες να παίρνουν το ρεύμα πιο φθηνά. Αυτό είναι αντικοινωνικό και είναι και ανεδαφικό και είναι και μη ρεαλιστικό. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, δεν θα πρέπει να εκπλησώμεθα που ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αυτή την αρνητική εικόνα και αυτή την απαξίωση. Ε, αν αυτά που είπατε εδώ βγείτε και τα πείτε πουθενά πιο έξω, δημόσια, στην κοινή γνώμη, θα μειωθεί κατακόρυφα η ε, δημοφιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει ε, να ε, βοηθάμε τους καταναλωτές και σε περίπτωση που το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάρα πολύ αδύνατο, να αξίζει τον κόπο να επενδύει κάποιος. Και όχι να έχουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Τσεχία ή στην Πολωνία να πρέπει να φτιάξουμε εμείς μετασχηματιστές για να μπορούμε να μεταφέρουμε το ρεύμα. Δεν το αναφέρατε καν. Μιλήσατε για την οικονομία της αγοράς, στην οποία θα παραδίδονται όλα αυτά, αλλά ε, είναι αντιφατικά αυτά που μας λέτε. Εμείς πάντα λαμβάνουμε υπόψη και κοινωνικά στοιχεία και κάνουμε τα πάντα ε, για να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό μου λείπει από τη μελέτη σας. Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν το αντιμετωπίσουμε, τότε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τη χείριστη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε μια λύση, να βοηθάμε τους πολίτες για να τους κερδίσουμε στο πλευρό μας. Παράδειγμα, αν δουλεύατε σε ένα εργοστάσιο και σας έλεγε κάποιος ε, κάτι τέτοιο και σας υπαγόρευε ποιος θα σας πουλάει το ρεύμα και μάλιστα να ελέγχετε και το συμβόλαιο πριν το υπογράψει, θα γινόταν έξαλλος. Σας ευχαριστώ κύριο Σέριξον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να συζητήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα αυτό, πώς μπορούμε να καταφέρουμε να ε, λειτουργεί αποτελεσματικά η ενεργειακή αγορά, τι πρέπει να αλλάξουμε. Και στο ηλεκτρικό δίκτυο και στις διασυνδέσεις, όπου φτάνουμε στα ίδια συμπεράσματα. Η Επιτροπή και συνολικά το Κοινοβούλιο, σχετικά με το στόχο που ετέθη από πέρσι το φινόπορο. Ε, θα έλεγα ότι εκεί θα ήταν σημαντικό να μην εξαγάγουμε άλλα συμπεράσματα, αλλά καλύτερα τώρα να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση κατά την οποία το ηλεκτρικό δίκτυο στην Ευρώπη θα είναι καλύτερα συνδεδεμένο Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε περισσότερες ανανεώσιμες στο σύστημα. Σημαντικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι συνδέσεις μεταξύ των χωρών, αλλά εντός των χωρών. Και εδώ φαίνεται η Γερμανία ως παράδειγμα. Ε, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προβλήματα στην Πολωνία και στην Τσεχία. διότι τα ανανεώσιμα της Γερμανίας πρέπει να περάσουν από αυτές τις χώρες και δεν πάνε νότια απευθείας μέσω Βαβαρίας λοιπά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε περιφερειακούς στόχους. Να μην εστιαζόμαστε μόνο στο συνολικό στόχο, αλλά και στη διαδικασία την επιμέρους. Ευχαριστούμε τον κύριο Έριξον. Αναφέρατε την ε, Τσεχία και εκεί είχαμε την πρόταση του κυρίου Ζέμαν, αν δεν κάνω λάθος. Παρακολουθείτε λοιπόν, όπως βλέπω. Έξοχα. Συνάδελφοι, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ζητάει το λόγο, δεν βλέπω. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω δύο ερωτήσεις δικές μου. μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή αγορά χονδρικής, λέει ο κύριος Μπούζεκ. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάποια προβλήματα με τους κώδικες μετάδοσης, μεταφοράς, μεταξύ των κρατών μελών. Πώς το βλέπετε αυτό. Διότι οι διαχειριστές μεταφοράς η συνεργασία μεταξύ των TSO είναι η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς, αλλά αυτό είχε καθοριστεί στα πλαίσια της τρίτης ενεργειακής δέσμης από το 2009, πριν από 7 χρόνια. Έχουμε λοιπόν μήπως ε, κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την συνεργασία μεταξύ των ε, διαχειριστών. Γιατί αυτό για μένα είναι ένα σημαντικό ζήτημα υλοποίησης της τρίτης ενεργειακής δέσμης. Είχα πει ήδη πριν από καιρό ότι υλοποιείται πολύ χειρότερα η ενεργειακή δέσμη παρά ο κανονισμός για την προμήθεια φυσικού αερίου που ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Επίσης, η ανανέωση του δυναμικού, τα CRM, αναφερθήκατε και στις ανανεώσιμες δεν λαμβάνουμε υπόψη το κόστος μεταφοράς στο δίκτυο στην περίπτωση των ανανεωσίμων. Και λέω, η ανταγωνιστικότητα εντός της αγοράς είναι πολύ δύσκολη υπό την έννοια αυτή. Διότι το κόστος μεταφοράς των ανανεωσίμων είναι πιο υψηλό από των συμβατικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν και τις τιμές, το κόστος μεταφορά στο δίκτυο. Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε τους μηχανισμούς στήριξης των ανεωσίμων από το 2020. Ή να έχουμε αντίστοιχους μηχανισμούς στήριξης σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό αν θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς θα εναρμονίσουμε λοιπόν τα εθνικά στήματα στήριξης. Και μια τρίτη ερώτηση. Λέτε ότι δεν πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές, να έχουμε ανταγωνισμό. Μάλιστα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τον υπόλοιπο κόσμο συστήματος που να μην έχει καμία ρύθμιση για την τιμή του φυσικού αερίου και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και η ερώτησή μου είναι, αυτό κάτι τέτοιο λειτουργεί, μας βοηθάει πραγματικά η απουσία ρύθμισης. Εγώ είμαι υπέρ του συνθήματός σας να μην ρυθμίζουμε. Αλλά έχετε απτά παραδείγματα συγκεκριμένα να μας δώσετε. Καλύτερα θα ήταν από μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να είναι από, την Βολιβία, από τη Βολιβία ή τον Μπαγκλαντές. Τι να σας πω δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν έχετε παράδειγμα καλοδεχούμενο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ε, πάω σε μία-μία τις ερωτήσεις. Καταρχάς κύριε Κόλισεκ, δεν ήταν ένας από τους στόχους μελέτης οι κοινωνικές στοιχές, αλλά είναι σημαντικό. Υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα, είναι αλήθεια, στα ζητήματα τιμολόγησης, στην συνολική τιμή της, τελική μάλλον τιμή της ενέργειας, ώστε να πάμε προς την κατεύθυνση της μη ρύθμισης. Εμείς εξετάσαμε την Ενεργειακή Ένωση στο σύνολό τη ως προς το πώς θα μπορούσε ιδανικά να λειτουργεί. Δηλαδή αν κανείς πράγματι θέλει να πάει προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού, αν θέλει να έχει περισσότερους προμηθευτές, τότε είναι καλύτερο να μην ρυθμίζει τις τιμές. Γιατί είναι, αν ρυθμίζει είναι πιο δύσκολο για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές. Αλλά βεβαίως χρειάζεται χρόνο μια τέτοια μετάβαση. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου, δεν το ακούμε. like to build. Ε, θέλετε, αν θέλετε να επεκτείνετε την εκεί πηγή, πρέπει να έχετε μια συμφωνία επί των τιμών. Πώς θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας άλλη πηγή Με την απουσία του precast ή οποιοδήποτε ρυθμίσεω, Θα, θα είμαστε λίγο χαμένοι εκεί. Κοιτάξτε, μπορούμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Και οι δύο έχουμε δουλέψει σε επιχειρήσεις ενέργειας, έχουμε συζητήσει για μεγάλες επενδύσεις σε μεγάλες εταιρείε για επενδύσεις ευρωπαϊκές. Εγώ και στην Πολωνία έχω εργαστεί, για παράδειγμα, και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι απαραίτητα αυτή η περίπτωση. Επενδυτικός μιλώντας, αν θέλω να αναπτύξω ένα σχέδιο επιχείρησης και να πάω προς την, ε, πάση περιπτώσει, την επιχειρηματική ανάπτυξη του συστήματος αυτού, τότε ναι, πρέπει να συζητήσω και για αυτό το θέμα. Εδώ όμως μιλούμε για την αύξηση, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, μπορούμε μετά το, στο διάλειμμα να έχουμε μια διμερή συζήτηση για να βρούμε. Δημερός λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα, ναι, αυτό έλεγα, δημερός. Για τους περιφερειακούς στόχους ε, έγινε ένα σχόλιο. Αν διατρέξετε το έγγραφο, θα δείτε ότι ένας ενδιάμεσος στόχος προς την αποτελεσματική ένωση είναι η περιφερειακή στόχη και τα περιφερειακά, περιφερειακά πρότυπα. Γιατί τις περισσότερες φορές χωρίζονται σε πέντε κομμάτια εντός της Ενιακής Ένωσης αυτά. Μερικά από τα κομμάτια εργάζονται καλά. Πρέπει να συνεργάζονται όλα μαζί. Και αυτό επίσης χρειάζεται χρόνο. Αλλά είναι ένα ενδιάμεσο βήμα που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και που είναι υλοποιήσιμο και η Κομισιόν το επεξεργάζεται. Έχουμε τακτικές συναντήσεις για το περιφερειακό επίπεδο και όπως το αναφέρατε κι εσείς η τρίτη δέσμη είναι του 2011, είναι ακόμα αρκετά πρόσφατη δηλαδή, γιατί χρειάζεται χρόνος ε, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να έχει αρμοδιότητες, μιλάω για την Acer, για την NSOE και NSOG, ε, χρειάζεται χρόνο για να είναι επιχειρησιακά έτοιμοι όλοι αυτοί. Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δει πρόοδο. Και έχουμε δει ότι συνεργάζονται διμερώς, συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη και τους διαχειριστές δικτύου και εδώ εν μέρει απαντώ και στη δική σας ερώτηση. Η Acer κάνει καλή δουλειά. Αλλά χρειάζεται χρόνος να συνδυάσει κανείς όλες τις ε, επιμέρους ε, τοποθετήσεις των διαφόρων TSO. Αυτά τα συζητούμε εδώ και 15-20 χρόνια. Και έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο Τώρα βλέπουμε και την οπτική γωνία των κρατών μελών όπου σταδιακά συνεργαζόμαστε όλο και στενότερα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε 3-5 χρόνια, είναι υψηλά τεχνικής φύσεως, είναι, υπάρχουν διάφορες, διάφορα επίπεδα περιπλοκότητας, χρειάζεται χρόνο. Αλλά αν δείτε που, που έχει φτάσει η ACR, η e και η NSOG μαζί με την Κομισιόν, και αν δείτε και τον πίνακα με τις ε, διασυνδέσεις με τους διαφόρους φορείς εντός της Ένωσης, επί των διαφόρων θεματικών, θα δείτε ότι έχουν προοδεύσει. Αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν ο Λουκ θέλει να προσθέσει κάτι επί των υπολείπων. Ναι, έγινε μια ανα... αναφορά στο face shifters. Αυτό είναι ένα τεχνικό πάρα πολύ ζήτημα, αλλά έχει τη σημασία και το ενδιαφέρον του να το απαντήσουμε ίσως. Ε, ε, μετατροπής βάσεις φάσεις ε, και είναι θέμα των διαχειριστών του δικτύου αυτό. Ε, είναι μια δυσκολία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ανώτερο του εθνικού. Και οι επενδύσεις να αποφασίζονται έτσι. Για να μεγιστοποιούμε και ε, τις ε, κοινωνικές ε, ωφέλειες. Δεν ξέρω στην Πολωνία τι έγινε, αλλά συνήθως ε, οι επενδύσεις γίνονται βάσει εθνικού συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας. Κανονικά θα πρέπει για να βελτιστοποιούνται και οι επιλογές επενδυτικές να γίνεται αυτό σε επίπεδο ανώτερο του εθνικού. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο για την ολοκλήρωση της αγοράς. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε δύο περιπτώσεις, ειδικά ε, σε αυτό το θέμα. Θέλω επίσης να τονίσω την ανάγκη ε, να συμπεριληφθούν και οι αγορές ημερήσεις, intraday δηλαδή, ε, κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη και την ολοκλήρωση ε, των ανανεωσίμων. Είναι οι ενδοημερείς στις λεγόμενες αγορές αυτές και ενδιαφέρουν και τους διαχειριστές ε, των δικτύων, τους TSO και τους ε, φορείς της αγοράς, τους εμπορικούς. Καταλαβαίνετε ότι ε, οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να κανονίζουν την πορεία τους, τις εμπορικές τους ε, συναλλαγές ε, και οι διαχειριστές του δικτύου μεταφοράς επίσης. Έτσι το σύστημα γίνεται πολύ πιο οικονομικό και μπορούν οι διάφορες αγορές και οι διάφοροι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς να τα αξιοποιούν αυτά και να τα εκμεταλλεύονται. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύου μεταφοράς, είναι σημαντικό να υπάρχει πιο περιφερειακή ε, συνεργασία και διαρθρωμένη. Υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βέλτιστες πρακτικές και παράδειγμα προσμίμηση για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τα βασικά καθήκοντα που θα μπορούσε να αναθέσει κάποιο σε ένα υπερεθνικό επίπεδο να εκχωρηθούν, δηλαδή είναι επενδύσει σε κύριο λόγο, διασυνοριακέ, ε, υπολογισμοί και κατανομή χωρητικότητα, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και επίση οι προμήθειε. οι διαγωνισμοί ε, ε, για την προμήθεια ενέργειας με εξοικονόμηση και των πόρων και των αποθεματικών ε, άλλα σχόλια. Ε, κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα ή ζήτημα. Τι θα γίνει μετά το 2020 και πώς θα επιδοτούνται οι ανανεώσιμες. Θα υπάρξει ανάγκη ένα σύστημα ε, ε, πληρωμής και επιβράβευσης. Το σημερινό δεν είναι βιώσιμο γιατί πέφτουν πολύ τιμές και δεν πρόκειται να επανέλθουν στην παρούσα συγκυρία και φάση. Στη Γερμανία υπάρχει μια μελέτη για ένα νέο μοντέλο αγοράς χωρίς οροφές στις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια βεβαιότητα και ένας κίνδυνος για τους επενδυτές και παραμένει υψηλό και δεν επενδύουν σε αυτό τον κλάδο. Άρα θα χρειαστεί ένας μηχανισμός που να αμείβεται η παραγωγή ε, ε, ρεύματος από τις ανανεώσιμες. Γιατί όταν σχεδιάζεις ένα σύστημα τέτοιο για την αγορά θα πρέπει να συμπεριλάβεις και τις ανανεώσιμες. Άρα θα χρειαστεί κάποια συμπληρωματική ε, ρύθμιση Θα δούμε ποιος είναι ο στόχος για το 2030. Θα είναι δεσμευτικό σε εθνικό επίπεδο, θα υπάρχει δυνατότητα ε, για πιο συντονισμένη προσέγγιση με λιγότερες τρευλωτικές ε, πολιτικές. Ε. Στη μελέτη αυτό δεν το έχουμε μελετήσει, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ένα τελικό σχόλιο για τη ρύθμιση των τιμών, τιμολόγηση. Οι τιμές του τελικού καταναλωτή λιανικής θα πρέπει να είναι πιο δυναμικές και να ε, ακολουθούν και τις τιμές χονδρικής. Σήμερα σε κάποια κρατημέλη δεν συνδέεται αυτό, ε, δηλαδή η τιμή της λιανικής με την τιμή της χονδρικής. Ε, για να υπάρξει λοιπόν μια αντίδραση, μια ανταπόκριση, θα πρέπει και οι τιμές λιανικής να ανακλούν την κατάσταση στην αγορά και να δίνουν κίνητρα. Και θα πρέπει και οι λιανικοί καταναλωτές να προσαρμόζουν την κατανάλωση στις ανάγκες και στην κατάσταση της αγοράς. Εξού και τα εφή e, δίκτυα, smart grids κτλ. Υπάρχει κανένα καλό παράδειγμα σχετικά, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που τη θέσατε. Καλώς. Παρακαλώ, κύριε Κόχλιτσεκ, να τα πείτε διμερώς με τον κύριο Ιβανούφελ και με τον κύριο Ράντε Μάκερς να τα βρείτε για τα ερωτήματα που είχατε να τους θέσετε. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ε, συντάκτες της μελέτης. Όπως είδατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση να σας κάνω. Επιπλέον συνεδρίαση της Επιτροπής μας. 9η Μαΐου, ε, που είναι και η ε, νίκη μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 7 με 9 το βράδυ. Δευτέρα, στο Στρασβούργο. 9η Μαΐου, στο Στρασβούργο, έκτακτη συνέδρια της Επιτροπής, επιπλέον 7 με το βράδυ. Ειδική συνεδρία. με συγκεκριμένο θέμα και κοινή με την Επιτροπή Πολιτισμού, Ήτρα δηλαδή και ΚΑΛΤ, βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού. Έχουμε συναρμοδιότητα για τις, ε, ε, την έκθεση για τις δημιουργικές ε, επιχειρήσεις, το δημιουργικό κλάδο της οικονομίας. Ο ε, κύριος Έλερ είναι ο δικός μας εισηγητής. Σημαντική λοιπόν πληροφορία για όλους σας. 9 Μαΐου συνεδρίαση. Ο κύριος Λάγκεν, πρόεδρε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο διαδικαστικά για τον κανονισμό. Στην περασμένη θητεία προσπαθήσαμε πέντε χρόνια να καταργήσουμε τις συνεδριάσεις Δευτέρα στο Στρασβούργο. Τώρα υπογείως και περιέργως ε, παρισφρίουν και επανέρχονται. Είναι δύσκολη απόφαση. Ξέρω ότι το υποστηρίζουν οι συντονιστές, παρόλα αυτά εγώ το θεωρώ λάθος. Διότι πρώτον, τη Δευτέρα, πολλοί συνάδελφοι φτάνουν στο Στρασβούργο, δεύτερον έχουμε ολομέλεια και τρίτον, ε, συνεδριάζουν και πολιτικές ομάδες προηγουμένως. Τώρα αν έχει αποφασιστεί τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά εσείς που είστε και πρόεδρος της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει στο μέλλον να φροντίσετε να μην το κάνουμε σύστημα κάθε Δευτέρα όσο φτάνει καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάγκεν θα μπορούσαμε ίσως να βάλουμε τη συνεδρίασή μας στις 8 αντί για τις 7. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα για σας. 8 με 10. Όχι. Α, δεν θέλετε καμία συνεδρίαση από ό,τι κατάλαβα. εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα. Βλέπετε όμως ότι είναι κάτι το απρόσμενο. γιατί έπρεπε να κάνουμε από κοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού και έτσι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Βάσει του κανόνα 55 πρέπει να υπάρξει κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών με τους δύο εισηγητές. Επομένω, δυστυχώ δεν υπήρξε διαφορετική δυνατότητα. Χρονικά δηλαδή δεν έβγαινε και για εμάς και για την Επιτροπή Πολιτισμού. Εάν υπήρχε μεγαλύτερη ευχαίρεια χρόνου, θα τα κάναμε διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά τώρα δεν γινόταν διαφορετικά, γι' αυτό προτείναμε μία επιπρόσθετη συνεδρίαση. Λυπάμαι, κύριε Λάγκεν, ούτε εμένα μ' αρέσουν αυτέ οι συνεδριάσει, αλλά συμφωνούμε ότι αυτή τη φορά είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Επαναρχόμαστε στι 3. Προς νέο σχεδιασμό της αγοράς. Ο κύριος Λάγκε θα περιμένει μέχρι τις 3. Εντάξει, είστε έτοιμος για όλα. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, συντάκτες της μελέτης. Ευχαριστώ και για την υπομονή σας που μείνατε μέχρι το τέλος.